Why don't we start? Uh, <laughs> I don't want to uh, uh, wait for the ones who are late. Να ξεκινήσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω στα γαλλικά. Ας μην περιμένουμε άλλο τους καθυστερημένους. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Να, ευχαριστώ να ευχαριστήσω τον Κρίς που με αντικατέστησε εχθές. Και να σας πω ότι ήμουν στη Γαλλία στην επέτειο, μάλλον στην εκδήλωση που έγινε για τους 13 νεκρούς στρατιωτικούς στην επιχείρηση Μπαρκάν στο Μαλί. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, ο πρόεδρος του Μαλί ήταν παρόν και αρκετοί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών Είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές όταν μιλούμε για θανάτους ε, στο πεδίο της μάχης αλλά και το, την σημασία της επιχείρησής τους ε, στο Σαχέλ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ε, του τζιχαντισμού η οποία κερδίζει έδαφος ιδιαίτερα στην Μπουρκίνα Φάσο. Έχουμε διάφορες αποστολές στο Μαλί, Μπαρκάν, UTM, Μίνουσμα και το G5 ε, στο Σαχέλ ε, προσπαθούν να σταθεροποιήσουν, να ομαλοποιήσουν την κατάσταση. Έχουμε άνω των χιλίων νεκρών και πάρα πολλούς εκτοπισμένους. Ε, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την ειρήνευση της περιοχής και την ασφάλεια τη δική τους και τη δική μας ε, υπάρχουν δυνητικά πολύ σημαντικές επιπτώσεις από τις συγκρούσεις αυτές. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα εθνικήνα που απέστειλαν δυνάμεις, ε, μάχημες ή όχι, στις αποστολές αυτές. Έχουμε και τη δύναμη κουμπά ειδική ευρωπαϊκή δύναμη που συνοδεύει τις ειδικέ αφρικανικές δυνάμεις που είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη θέση μας όταν έχουμε τέτοιου είδους συγκρούσεις που δεν, είναι καθόλου, που δεν χρησιμοποιούν καθόλου παραδοσιακές μεθόδους. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε και αποτυχίες, είναι μακρόπροθεσμη προσπάθεια. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. και για την προπαρασκευή, για την έρευνα στα αμυντικά θέματα. Να ευχαριστήσω την κυρία Κάιντς Χούμπερ στην ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και ε, τον εκπρόσωπο της, ε, του Οργανισμού Αμήνης που θα μας μιλήσουν για τα θέματα ερεύνης ε, στα, στην άμυνα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμέκ για την ε, αποστολή επίσκεψης 18 ε, Νοεμβρίου. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να παραστώ, αλλά μου είπαν, έμαθα, ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. 12 Νοεμβρίου το Συμβούλιο υιοθέτησε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού για το 2020, χαιρέτησε τη συνεισφορά του οργανισμού για την συνδιοργάνωση διαφόρων πρωτοβουλειών αμήνης αμυντικών θεμάτων. Έχουμε και τον διευθυντή EDIDP για να το πω σε καλά γαλλικά λέει πρόεδρος. Και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε και το Ταμείο Αμήνης. Στα πλαίσια της αξιολόγηση του, αυτής της PADR, της προπαρασκευαστικής αυτής δράσης και να αναπτύξουμε τις δυνατότητες που θα χρειαζόμαστε ώστε να υποστηρίξουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα τα πολιτικά θέματα εκτός των αμυντικών. Ήταν μια πρώτη σημαντική φάση το PADR για να εκδηλωθεί η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ για το 2019 και η φιλοδοξία είναι να ενισχυθεί η συνεργασία στα αμυντικά θέματα. Ο οργανισμός ε, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και σας δίνω το λόγο για 15 λεπτά περίπου, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να συνομιλήσω μαζί σας για το πιλωτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση. Θα γνωρίζετε ότι η στρατηγική ενέχει μια σειρά από πρωτοβουλίες που αλλάζουν το τοπίο, το αμυντικό και της ερεύνης στα θέματα αμήνης. Στο πλαίσιο των δύο αυτών προγραμμάτων προετοιμάζουμε το έδαφος για μια ισχυρή διάσταση ερεύνης στα αμυντικά θέματα στα πλαίσια του επομένου ΠΔΠ. Θα θυμάστε ίσως ότι το πιλωτικό είχε εισαχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό 15 και 16 προκειμένου να δοκιμάσουμε την πιο αποτελεσματική χρήση πόρων αμυντικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του προϋπολογισμού από τον EDA. Έγινε μια συμφωνία εξουσιοδότησης το Νοέμβριο του 2015 και ο οργανισμός κατέστη υπεύθυνο για την διαχείριση του πολιτικού προγράμματος και των δράσεων υπό αυτό. Αυτά έγιναν με έναν πολύ μικρό προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια, αλλά ήταν μια καλή αρχή της πρωτοβουλίας στα θέματα αμήνης και με χαρά μπορώ να σας πω πλέον ότι και οι τρεις πιλωτικές δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και όλες οι συνδεδεμένες δραστηριότητες υπό την εξοδότηση στο πρώτο εξάμεινο του 2019. Είναι ένα πλαίσιο ευκαιρίας να δοκιμάσουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με την βιομηχανία, τον κλάδο για τα θέματα αμυντικής ερεύνης. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υποεπιτροπή που είναι από την αρχή της προσπάθειας αυτής, της πρωτοβουλίας και μας παρέχει ένα πρώτο πλαίσιο, ένα πρώτο μορφότυπο. Προετοιμάζουμε εδώ το έδαφος και για την εκκίνηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την αμυντική έρευνα με 19 εκατομμύρια ευρώ σε τρία έτη. Η δράση αυτή είναι πολύ ευρύτερης κλίμακος από το πρόγραμμα και ξεκίνησε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία της αμυντικής έρευνας. Πρόκειται λοιπόν για μια γενικευμένη δοκιμή για να αποδείξουμε τη σημασία της έρευνας στα θέματα αυτά και για να θεμελιώσουμε την αμυντική μας συνεργασία. Και εδώ είχαμε μια συμφωνία αξιοδότησης το Μάιο του 2017 η οποία προβλέπει διαχειριστική αμοιβή για το κόστος που άμεσα συνδέεται με την υλοποίηση μέχρι το 5% και πέραν αυτού το πρόγραμμα υποφελείται από την εμπειρογνωμοσύνη του EDA στα θέματα αμυντικής έρευνας προκειμένου να υποστηρίξει τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματική παρακολούθηση των δράσεων. Συμπεριλαμβάνονται τρία προγράμματα εργασία σε τρία έτη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Ο εγκεκριμένο προπολογισμό ήταν 25 εκατομμύρια για το 2017, 40 για το 2018 και 5 για το 19. Αυτό το σύνολο το 90 μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε διάφορα εργαλεία και διάφορες δράσεις ερεύνης ώστε να έχουμε μια παραγωγική διάσταση αμυντικής έρευνας στο μέλλον. Συνολικά, έχουμε οδηγηθεί σε αυτά αποτελέσματα στις περιοχές που είχαν προηγουμένως ταυτοποιηθεί. με τις προπαρασκευαστικές δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα έχουμε πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις οι εκθέσεις των ε, ανεξαρτήτων παρατηρητών επίσης υπήρξαν θετικές να σας δώσω τώρα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις αυτές στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας του ΚΑΕΠΤΑ είχαμε 24 προτάσεις υπευλήθησαν δηλαδή και τα χρηματοδοτικά προγράμματα ήταν για τεχνολογικά συστήματα θαλάσσια, ε, προκεχωρημένα συστήματα ε, στρατού ξηράς. Μετά ε, λάβαμε οκτώ προτάσεις, το επόμενο έτος, το 18, για laser effectors, και συστήματα ε, ηλεκτρονικών ε, ε, τέλος πάντων ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία προγράμματα συμμετείχαν οντότητες από 26 χώρες. Το 2017 είχαμε το 41% των συμμετεχομένων στις συμπράξεις που ήταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 27% άλλους συμμετέχοντες και 17% ερευνητικά κέντρα. Το οποίο εξελίχθηκε σε 19% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 27% ε, αν ακούσαμε καλά τον ομιλητή για ερευνητικά κέντρα. Είχαμε ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ως επόμενες θεματικές ε, και συστήματα μη επανδρομένα περιοχές όπως η τεχνητή νοημοσύνη για τα θέματα τα αμυντικά, η τεχνολογία quantum και συστήματα ε, χρονισμού και και πλοήγησης. Ε, έχουμε η αξιολόγηση των προτάσεων των τελευταίων που λάβαμε ε, τρέχει ακόμα και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε αρχές του επόμενου έτους για τα διδάγματα που έχουμε μέχρι εδώ. Επιτρέψτε μου κάποιες συγκεκριμένε παρατηρήσεις. τις οποίες συντάξαμε από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας για το μέλλον, για την διαμόρφωση του αμυντικού ταμείου. Δοκιμάζοντας συνεργασία λοιπόν μεταξύ του EDA και τη Επιτροπή προκύπτουν κάποιες μέθοδοι σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Δοκιμάζουμε και τις ειδικέ εκθέσεις που υποβάλλονται. Τα ρυθμιστικά θέματα των δικαιωμάτων θα πρέπει να πετυχαίνουν μια ισορροπία μεταξύ της ομαλής ροής πληροφοριών και της προστασίας των πληροφοριών που παράγεται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντας ότι τα Υπουργεία Μήνης που είναι οι τελικοί χρήστες των τεχνολογιών θα έχουν επαρκή δικαιώματα πρόσβασης, λέει ο μελητή. Δοκιμάσαμε επίσης τρόπους που μπορούμε να διαβουλευόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς, πώς να διαμορφώνουμε καλύτερα τις θεματικές και πώς θα λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες της αμυντικής και τις ανάγκες. Πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, στις περιγραφές των θεμάτων τις ε, δραστηριότητες της συνδεδεμένες και παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, γιατί η ανάπτυξη βιωσίμων συστημάτων χωρίς επαρκές τεχνικές προδιαγραφές, που δεν θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεών μας, θα ήταν κατασπατάλες του δημοσίου χρήματος. Για τον EBA, βλέπουμε ότι ο ρόλος του μπορεί να είναι τριπλός να συμπεριλαμβάνει, μάλλον να διέπει τη διαδικασία υλοποίηση τη δραστηριότητε downstream αλλά και upstream, λέει ο Δηλαδή, upstream. Η υποστήριξη των κρατών μελών και τη Επιτροπή στην προετοιμασία του προγράμματο εργασία επί τη βάση των εργαλείων προτεραιοποίηση του EDA. Υλοποίηση και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέθεσε τις δύο, τα δύο πλαίσια δευτεριότητα στον EDA υπό εξοδότηση από την εκκίνηση, την υποβολή δηλαδή των προτάσεων, μέχρι την υλοποίηση. Το downstream είναι η καλύτερη ενσωμάτωση, αν θέλετε, ε, των ε, πορισμάτων της έρευνας στη δραστηριότητα αυτή. Υποστηρίζουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διαμόρφωση της δράσης αυτής, ε, συναντήσεις συντονισμού με τα κράτη-μέλη, ε, εξέταση θεμάτων που έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη, καλύτερη προτεραιοποίηση, καλύτερο clustering, λέει ο μιλητής, και ίσως πιο συγκεκριμένη εξέταση των θεματικών. Επίσης έχουμε το συνολικό στρατηγικό θεματολόγιο που θα διαμορφώσει την, το μελλοντικό πρόγραμμα εργασία του EDF του Ταμείου. Όπως λέει και ο πρόταση κανονισμού του. Επίσης έχουμε μία διάσταση ερευνητική στα πλαίσια του Ταμείου αυτού, που και εδώ όμως θα πρέπει να δούμε ξεχωριστούς τομείς ε, χρηματοδότησης, ε, στους οποίους συμβάλλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας βάσει συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική η ζήτηση, αλλά και οι αμυντικές επενδύσεις από τα κράτη-μέλη. Επομένως, θα πρέπει να αποφύγουμε εδώ πέρα αλληλοεπικαλύψεις όσον αφορά την έρευνα και τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό τα πιλωτικά προγράμματα και η προπαρασκευαστική δράση να έχουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση και έχουμε δει μέχρι στιγμή ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα μπορεί πραγματικά να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά όλη την εφαρμογή των πιλωτικών αυτών προγραμμάτων. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα μπορεί να συλλέξει του απαραίτητου πόρου που απαιτούνται προκειμένου να επιτελεστούν όλε αυτέ οι ερευνητικέ δραστηριότητε. Όσον αφορά τώρα την πρακτική εφαρμογή, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι το αρχικό σκεπτικό και αρχική στόχη τόσο των πιλωτικών προγραμμάτων αλλά και τη προπαραβαστική δράση έχουν επιτευχθεί, επομένως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να ανταποκριθεί στι ερευνητικέ ανάγκε όσον αφορά τον τομέα τη Άμυνα. Όσον αφορά τώρα τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της δράσης, τα δύο πρώτα προγράμματα εργασίας έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εξελίχθηκαν θετικά, δεχθήκαμε προτάσεις, έγιναν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμφωνίες, σε επιλέξιμα μάλλον προγράμματα, τα οποία κατέληξαν σε συμφωνίες εφαρμογής τόσο και το 2017 και το 2018. Περιμένουμε να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή ε, επεξεργαζόμαστε τις ε, υπόλοιπες επιλέξιμες προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε πώς ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να εκμεταλλευτούν και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα αυτά της έρευνας που λαμβάνει η χώρα σε κοινοτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένα προγράμματα follow-on, παρακολούθησης, ε, συνέχισης, ε, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ή σε εθνικό επίπεδο ή σε διμερές επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να μεταφράσουν την έρευνα αυτή σε μελλοντικέ στρατιωτικέ ικανότητε και δυνατότητε. Μόνο αυτό θα κάνει την αμυντική μα βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, καλύπτοντα τι στρατιωτικέ ανάγκε των ενόπλων δυνάμεών μα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όσον αφορά το Pilot Project Eurosmall, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και τα κράτη, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να υποφελούνται από το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα τεχνικά προβλήματα και να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά την έρευνα αυτή που έχει επιτελεστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρω... Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ιεραρχήσει τους ερευνητικούς πρωταρχικούς τομείς και αυτοί διαφαίνονται πλέον και στο πρόγραμμα εργασία το οποίο έχει εκπονήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά η ερευνητική μα δραστηριότητα να ανταποκρίνεται στι πραγματικέ αμυντικέ ανάγκε των κρατών μελών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας λοιπόν έχει εφαρμόσει σε όλα τα στάδια, του αρχικό και το μεταγενέστερο στάδιο, όλες τις φάσεις του ερευνητικού αυτού προγράμματος. Και όλοι οι δείκτες που έχουμε στα χέρια μας καταδεικνύουν ότι η ερευνητική μας δραστηριότητα είναι όντω αποτελεσματική και παραγωγική. Βάσει τώρα της προπαρασκευαστικής δράσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να συμβάλλουν με εθνικά προγράμματα στο Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα έρευνα στον τομέα της άμυνας. Βάσει αποφάσεων του Steering Board του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας υποβάλλουμε έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εκπονηθεί ένας αρχικός οδικός χάρτης για το ερευνητικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας. Τα κράτη-μέλη καταλήγουν σε ένα κοινό κείμενο το οποίο ιεραρχεί τις βασικές ερευνητικές προτεραιότητες των κρατών μελών, τις βασικές αμυνικές τους ανάγκες, καθώς επίσης και τους τομείς εκείνους στους οποίους υπάρχει ήδη μία συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Μέσω του εγγράφου αυτού, του οδικού χάρτη δηλαδή, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τόσο τη θεωρητική έρευνα που επιτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και την πρακτική εφαρμοσμένη έρευνα που έχει γίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε από κοινού κράτη-μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση στους βασικούς ερευνητικούς στόχους. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν τώρα να ζητήσουν από, την από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να συμβάλλει στην υποβολή ενός εγγράφου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις ε, ερευνητικέ αμυντικές ανάγκες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από πρωτοβουλία των κρατών μελών, η EDA έχει δημιουργήσει ένα άτυπο φόρουμ, το οποίο θα δημιουργήσει ουσιαστικά έναν χώρο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, καθώς επίσης και του EDIDP, του προγράμματος μηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν εν συνεχεία να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Ένα σημαντικό επίτευγμά μα επίση είναι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω των πιλωτικών προγραμμάτων και τη προπαρασκευαστική δράση επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο πλευρέ είναι προσιλωμένε στην κοινή συνεργασία προκειμένου να στεφτεί με επιτυχία η ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Άμυνα. Ευθυγραμμίζουμε την εργασία μας με αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα χαρακτηρίσει και οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία σε οποιονδήποτε ερευνητικό τομέα. Με την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν και οι δύο πλευρέ, τόσο ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, όσο βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη που υπάρχει από διάφορου τομεί στην ευρωπαϊκή αγορά, έχουμε πλέον τι απαραίτητε δεξιότητε που είναι απαραίτητε προκειμένου να στεφτούν με επιτυχία τόσο η προπαρασκευαστική δράση όσο και τα πιλωτικά προγράμματα. Εν κατακλείδη θεωρώ ότι οι προπαρασκευαστικές ε, δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα έχουν ε, αποτελέσει μια πολύ επιτυχή δοκιμή όσον αφορά την ερευνητική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία η οποία είναι ανταγωνιστική, η οποία να συνεργάζεται και κατά αυτόν τον τρόπο να καλύπτει τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αμυντική έρευνα και του αμυντικού εξοπλισμού. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα έχει πλέον την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να υποστηρίξει την όλη αυτή εργασία στα αρχικά, πρωταρχικά τη στάδια αλλά και στα μεταγενέστερα στάδια. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με έναν ε, γενικότερο σκεπτικισμό, ο οποίο ήταν διάχυτο πριν από μερικά χρόνια, όσον αφορά τις ικανότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και την προπαρασκευαστική δράση. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ε, Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας να σας ε, ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να ευχαριστήσω βέβαια και τον συνάδελφο από, την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που είχε καλύψει βέβαια τα περισσότερα ζημία τα οποία θα ήθελα να καλύψω. Όσον αφορά το ζήτημα της συνεργασίας ε, που ήταν ένα σημαντικό σημείο της Προπαρασκευαστική δράση. Μέσω τη συνεργασία αυτή, προσπαθήσαμε πραγματικά να δούμε ποιου μηχανισμού θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν και μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να δούμε πώς θα καταφέρναμε να χρηματοδοτήσουμε για πρώτη φορά την ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ευρωπαϊκά κονδύλια και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. και προσπαθήσαμε να δούμε στον τομέα αυτό πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ο Χόρκε αναφέρθηκε στην κατανομή αυτή των καθηκόντων που θα μπορούσαμε να είχαμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αυτό φάνηκε μέσω της προπαρασκευαστικής δράσης και μέσω των πιλωτικών προγραμμάτων που αποτελούν ένα πρώτο δείγμα της πλήρους σφαιρικής συνεργασίας που θα μπορούσαμε να είχαμε μεταξύ των δύο αυτών οργάνων στο μέλλον, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Προχωρήσαμε σε προσκλήση υποβολής προτάσεων, δεχθήκαμε τις ερευνητικές προτάσεις, τις ερευνητικές προσφορές από τα κράτη-μέλη και προσπαθήσαμε έπειτα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα το οποίο μοιάζει με αυτό της επιτροπολογίας να δούμε ποια προγράμματα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως επιλέξιμα και ποια τελικά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο μέλλον. Και κατά αυτόν τον τρόπο εκπροσωπήθηκαν και τα κράτη-μέλη σε έναν καινοτόμο τρόπο εργασίας. Αυτή τη στιγμή στετήσια προγράμματα εργασίας θεσπίστηκαν Είχαμε και το νοδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσαρτήθηκε σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας και έπειτα κληθήκαμε να προχωρήσουμε στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και να κάνουμε τις απαραίτητες αξιολογήσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ξέρετε ότι αυτό είναι ο συνήθις τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιλογή ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό θα κάναμε και για τα μη στρατιωτικά προγράμματα. Ο Χόρκε αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα της παρακολούθησης, της επιτήρησης των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων που έγινε και η επιτήρηση αυτή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης είχαμε και έλεγχο δεοντολογικής φύσης των προτάσεων που υποβλήθηκαν. Και στη συνέχεια είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ο οποίος μέσω της συμφωνίας αυτής ανάθεσης αρμοδιοτήτων ασχολήθηκε με την όλη διαδικασία μετά την επιλογή και την αξιολόγηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Πού βρισκόμαστε τώρα επί του παρόντος. Σας μην επαναλάβω όλα τα αριθμητικά δεδομένα που σας έδωσε πριν από λίγο ο Χόρχε, Πάντως όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αντλήσουμε συγκεκριμένα διδάγματα από την προπαρασκευαστική αυτή δράση ως προς τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να είχαν τα ερευνητικά αυτά προγράμματα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το οποίο θέλαμε να δοκιμάσουμε είναι πώς λειτουργούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί πώς θα μπορούσαμε ουσιαστικά να συντονίσουμε και να οργανώσουμε την ε, αμυντική έρευνα, αυτή δηλαδή η οποία ανταποκρίνεται στις πραγματικές στρατιωτικές ανάγκες και απαιτήσει. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα είδος έρευνα το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί από το συμβατικό ε, πλαίσιο έρευνα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δηλαδή το οποίο ασχολείται με τους μη στρατιωτικού τομεί. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες πτυχές στον τομέα αυτών τη έρευνα, τις οποίες κρίναμε ως θετικές. Τώρα υπήρχε πραγματικά έρευνα από την αμυντική κοινότητα. Μπορούμε σαφώς να δώσουμε εδώ μια καταφατική απάντηση. Σαφώς υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον. ανεφέρθηκε σε αυτό και, το, σε αυτό και ο Χόρχε. Είχαμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και φάνηκε αυτό και από το έντονο ενδιαφέρον το οποίο υπήρξε στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Μόνο και μόνο το 2019 είχαμε 94 συνολικά προτάσεις που υπευλήθησαν και οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή 10 συμβάσεων και φέτος, μόνο και μόνο φέτος, δηλαδή το 2019. Τώρα, η προπαρασκευαστική λοιπόν δράση οδήγησε πραγματικά στην ανταπόκριση που θέλαμε. Θα έλεγα ναι. Ήταν πολύ θετική και ενθαρρυντική ανταπόκριση και είδαμε ότι αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η προπαρασκευαστική δράση, κινητοποιήθηκαν αρκετά κράτη-μέλη προκειμένου να συμβάλλουν σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Είχαμε λοιπόν καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μάλιστα πολλές φορές ήταν και διασυνοριακή. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ανταπόκρισης που είχαμε είναι ιδιαίτερα θετικά. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θελήσαμε να εξετάσουμε είναι να δούμε αν αυτή η προπαρασκευαστική δράση και αν τα ερευνητικά αυτά προγράμματα πραγματικά κινητοποίησαν όλα τα κράτη-μέλη, αν δόθηκαν οι ευκαιρίε σε όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Ακούστηκαν εν αρχή κάποιε επικρίσει. Ορισμένοι είπαν ότι ε, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στα συνήθι μεγάλα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα και που έχουν ήδη μια παγιωμένη αμυντική βιομηχανία. Μέχρι στιγμή στι προτάσει που λάβαμε, αλλά και στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε μέσω της προπαρασκευαστικής δράσης τα τελευταία δύο χρόνια, 26 κράτη-μέλη σε σύνολο 28 εκπροσωπούνται είτε μέσω της ίδιας της βιομηχανίας, είτε μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε μέσω συμμετοχής στις ε, διάφορες κοινοπραξίες. Επίσης, εφαρμόζοντας την προπαρασκευαστική δράση, θέλαμε να δούμε πόσο συμμετέχουν και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματικά μπορούμε να προσελκύσουμε στα ερευνητικά αυτά προγράμματα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τα 7 ερευνητικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, είχαμε, είδαμε ότι από τους 106 δικαιούχους, οι 24 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δύσκολο βέβαια είναι να δει πραγματικά κανείς ποιες επιχειρήσεις είναι όντω μικρομεσαίες. Αν δούμε όμως τα, τα, στατιστικά δεδομένα βλέπουμε ότι έχουμε μια συμμετοχή της τάξης του 23% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την προπαρασκευαστική δράση και ένα 11% από τον διαθέσιμο προπολογισμό μας πηγαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάλι όμως αυτό εξαρτάται από το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό καθεαυτό όπου βλέπουμε ότι ανάλογα με το πρόγραμμα ένα 2 με 48% του προπολογισμού δίνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προέρχονται από 10 διαφορετικά κράτη-μέλη και συμμετέχουν στις κοινοπραξίες αυτές. Και έχουμε κυρίως εκπροσώπηση από την Ιταλία, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά όμως αποτελούν θετικό αποτέλεσμα της προπαρασκευαστικής δράσης. Δεν ελήφθη καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκειμένου να προωθηθούν ή να ευνοηθούν αναγκαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται πλέον αυτή τη στιγμή όπου έχουμε συγκεκριμένους μηχανισμούς για να προωθήσουμε περισσότερο τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τον αρχικό μας προπολογισμό, όταν είχαμε δηλαδή μόνο 90 εκατομμύρια, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ευνοήσουμε συγκεκριμένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, το ζήτημα της ε, ανάθεσης, το ζήτημα των ε, επιδοτήσεων. Εδώ πέρα προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις συνθήκες οι οποίες πραγματικά προβλέπονται στην ε, σύναψη των συμφωνιών και μέσα σε 9 μήνες προσπαθούμε να προχωρήσουμε στην ανάθεση και τη χρηματοδότηση των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων σε συγκεκριμένε επιχειρήσει. Θα έλεγα ότι τα συμπεράσματα που έχουμε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Έχει στεφθεί με επιτυχία η προπαρασκευαστική δράση και τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε είναι σίγουρα θετικά και ελπιδοφόρα. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον. Μέσω της εφαρμογής της ε, προπαρασκευαστικής δράσης ε, ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εντοπίσει κάποια θετικά στοιχεία όσον αφορά την πολιτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Εμείς προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε κανόνες για την αμυντική έρευνα, οι οποίοι μοιάζουν τελικά με τους κανόνες που έχουμε ήδη για την έρευνα στον τομέα των μη στρατιωτικό, προσπαθώντας βέβαια να τηρήσουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει ο αμυντικός τομέας. Οι, οι κανόνες αυτοί λοιπόν που εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη θα πρέπει τώρα να εφαρμοστούν και στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο από το 2021 θα συνδυάζει τόσο την πτυχή της έρευνας όσο και την πτυχή που έχει να κάνει με τις ε, αμυντικές δυνατότητες και ικανότητες και που θα συνδυάζεται πλέον με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας. Οι κανόνε αυτοί λοιπόν που εφαρμόσαμε στην προπαρασκευαστική δράση και που πέρασαν έπειτα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο σύστημα υποβολή αναφορών όπου τα κράτη-μέλη πέρα από τι ε, τακτικέ αναφορέ που υποβάλλουν και στον τομέα τη ε, μη στρατιωτική έρευνα. είναι πολύ σημαντικό να υποβάλλουν και εκθέσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των ε, προγραμμάτων των ερευνητικών που χρηματοδοτούνται από την προπαρασκευαστική δράση και στόχος μας είναι κάθε φορά να διασφαλίζουμε ότι οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες δεν θα είναι μόνο θεωρητικές, δεν θα καταλήγουν ε, τελικά να μην εφαρμόζονται, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δρομολογούν ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει εν συνεχεία να μπορούν να έχουν και πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα των κοινοπραξιών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έπειτα και μία έκθεση follow-up που να δείχνει πώς στην πράξη εφαρμόστηκε η έρευνα, πώς έδωσε δηλαδή χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό δηλαδή, αυτός είναι ένας νέος κανόνας που έχουμε εντάξει στην προπαρασκευαστική δράση. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Θα συνεχιστούν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν και κάποιοι νέοι διαφορετικοί κανόνες που έχουν να κάνουν κυρίως με το στάδιο της εφαρμογής, ενώ στην προπαρασκευαστική δράση είχαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ως βασικό εταίρο, Τώρα στα πλαίσια του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης τομέα της άμυνας δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ρόλο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα και στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα δεν προβλέπεται αυτή η υποχρέωση όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Υποχρέωση η οποία περνάει τώρα στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το οποίο θα χρηματοδοτείται από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πέτρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύ πλήρες εξηγήσεις. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να διασαφηνίσουμε κάποια σημεία. Έχουμε από το 17 και 18 κάποια διδάγματα μετά από τους διαγωνισμούς που οργανώθηκαν. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που ουσιαστικά αφήνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός της συμμετοχής ε, σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Υπάρχουν γενικοί λόγοι που εξηγούν αυτή την, ε, τον αποκλεισμό, είτε είναι κάτι που εξαρτάται από τη χώρα. Δεύτερη ερώτηση, ποιος παίρνει την απόφαση όσον αφορά τις προτεραιότητες που τίθενται για το ερευνητικό πρόγραμμα του κάθε Ποιος είναι ο οργανισμός, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της εξωτερικής πολιτικής, αυτές οι προτεραιότητες κατά κάποιο τρόπο συντονίζονται. Υπάρχει δηλαδή ε, ένα συντονισμό των προτεραιοτήτων σε κάποια στάδια αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ πλήρης η παρουσιάση σας και από ό,τι καταλαβαίνω πραγματικά προσπαθήστε να ξεπεράσετε αυτόν τον κατακαιρματισμό όσον αφορά τα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της άμυνας. Σήμερα γίνεται η μεγάλη συνάντηση κορυφής ε, του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και όλες οι τελευταίες ε, συναντήσεις κορυφής του ΝΑΤΟ είχαν ε, σαν θέμα το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι δαπανούν αρκετά κονδύλια για την άμυνα και είναι η μόνιμη, αν θέλετε, κριτική από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς μπορούμε εδώ να αξιοποιήσουμε καλύτερα ενδεχομένως τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται. Πώς μπορούμε να είμαστε στο επίπεδο των συμμάχων μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Αρκεί αυτό που δαπανούμε όταν μιλάμε για εξοπλιστικά προγράμματα, για το θέμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και της ε, κυριαρχίας της Ευρώπης. Είμαστε σε πολλούς από αυτούς τους τομείς αρκετά πίσω. Τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κρίς Πέτρας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι το ίδιο θέμα που έθεσε και ο συνάδελφος. Εχθές αναφερθήκαμε στα προγράμματα ανάπτυξης ε, της αμυντικής ε, και εξοπλιστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Και εχθές ακούσαμε ότι η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν ξεπνάει το 11%. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις 33%. Δεν λέω ότι είναι μικρό το ποσοστό το 33%, αλλά πώς μπορούμε να το αυξήσουμε. Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος, υπάρχει η πρωτοβουλία αυτή την οποία συζητάμε σήμερα, αλλά και πολλές άλλες. Υπάρχει συντονισμός, υπάρχει κοινή επιλογή προτεραιοτήτων, έτσι ώστε να αποφύγουμε επικαλύψεις. Τρίτον, σήμερα υπάρχει η μεγάλη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και καταλαβαίνω ότι το θέμα του διαστήματος θα συζητηθεί και θα υπάρξει μία επίσημη δήλωση των ηγετών στα πλαίσια αυτής της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ για το διάστημα, το διάστημα το οποίο θα ορίζεται πλέον σαν πεδίο επιχειρήσεων. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς βλέπετε εσείς αυτή την πολύ σημαντική απόφαση που σίγουρα θα ληφθεί σήμερα ή αύριο. Τράιν Μπασέσκου για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας παρουσιάσατε. Ακούγοντάς σας, πολύ ειλικρινά, ε, μου έρχεται μια σκέψη. Επενδύουμε πολύ λίγο, πολύ χαμηλά ποσά. Όλοι περιμένουν τεράστια αποτελέσματα, ενώ τα ποσά που επενδύουμε είναι ελάχιστα. Εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό τομέα, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να συνεργαστούν, να συνδυάσουν τη χρηματοδότησή τους με καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν στον τομέα της έρευνας. Κοιτάξτε τι κάνουμε στην πράξη, στην εξοπλιστική βιομηχανία. Κοιτάξτε τη Ρουμανία και την Πολωνία παραδείγματος χάρη. Αγοράζουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, τα οπλικά μας συστήματα. Γιατί? Γιατί είναι πολύ απαρχαιωμένα τα ευρωπαϊκά συστήματα και έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις. Παραδείγματο χάρη, η πύραυλη Patriot για την ε, προστασία ένα σύστημα το οποίο αγοράζουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν υπάρχει αντίστοιχο οπλικό σύστημα αεράμινας στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχουν πέντε ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν παραγγείλει αεροσκάφη F-35 αντί να επιλέξουν τα Ραφάλ που είναι ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη. Γιατί το κάνουν αυτό. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει πραγματικά να δούμε πού βασίζονται αυτές οι επιλογές και να πάρουμε αποφάσεις καλύτερη συνεργασία στη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να αναπτύξουμε και να παράγουμε συστήματα αποτελεσματικά, πιο αποτελεσματικά, για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά με τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Οι συζητήσεις ε, όσον αφορά την απόδοση της εξοπλιστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη είναι πολλές, αλλά τελικά βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα της απόδοσης δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Δεν είμαστε στο καλύτερο επίπεδο. Πρόεδρος, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτά που λέτε υποστηρίζονται από τα περισσότερα μέλη αυτής της Επιτροπής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δικαίωμα να έχετε αυτή την άποψη. Κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο τμήμα του εξοπλισμού της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας ε, πηγαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια δεν λέω ότι τα αμερικανικά συστήματα τα πάνε άσχημα. Τώρα, η σημασία των πρωτοβουλίων ε, PADR είναι σημαντικό να μην συμμετέχουν επιχειρήσεις από κάποιες μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή επιχειρήσεων ή φορέων από μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τι είδους κατανομή δηλαδή έχουμε. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα προσέθετα και εγώ το εξή ερώτημα γιατί αναφερθήκατε στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα. Ε, θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε ένα μέγεθος, ένα ποσοστό που να εκφράζει την συμμετοχή των επιχειρήσεων ή εν πάση περιπτώσει τη βρετανική συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Thank you. Thank you for your, your questions. Um, Mr. Otrovicius, when you talk about, um, I think... Κοιτάξτε, και οι δύο παρουσιάσεις μας και τη Σιλβεκή δικιά μου δεν uh, παρουσίασαν ε, τους λόγους ή δεν είδαν ε, ποια, ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι μιας ε, μη επαρκούς συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Αντίθετα, θεωρούμε ότι σε όλους τους τομείς, σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ερευνητικό τομέα έχουν μία συμμετοχή που ξεπερνάει την παλιά πρακτική τους. Γιατί η έρευνα που γίνεται στην Ευρώπη έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο και οι προπολογισμοί που χρηματοδοτούν την έρευνα. Εξού και πολλές ε, από αυτές τις ε, επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται πλέον από εθνικούς πόρους. Αυτό λοιπόν υποχρέωσε πολλές από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εθνικά του σύνορα και να λειτουργήσουν ε, υπερεθνικά. Η Σίλβια σας είπε ότι θα υπάρξουν πλέον στα Ευρωπαϊκά Ταμεία κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ε, επαρκή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εργασιών αποφασίζεται από την Επιτροπή ΑΣΕΦ αυτό που κάναμε εμείς στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό από κοινού με τα κράτη-μέλη και βάσει βεβαίως του σχεδίου ανάπτυξης των δυνατοτήτων μπορέσαμε να εγγυηθούμε αν θέλετε μια συμμετοχή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα προγράμματα αυτά. Τώρα, πώς αυτό μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται με την ΠΕΣΚΟ και πώς συνδέεται αυτό ουσιαστικά με τις προτεραιότητες οι οποίες θα έπρεπε να είναι κοινέ. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία 25 ετών, 25 κρατών, συγγνώμη, για μια πιο συνεκτική πολιτική στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και έρευνας και τα περισσότερα προγράμματα σίγουρα ανταποκρίνονται και σε κοινά προγράμματα με την ΠΕΣΚΟ. Παρόλο που αυτά στοχεύουν πολύ περισσότερο ε, τις δυνατότητες. Παρόλα αυτά πολλές φορές η έρευνα είναι κοινή. Και βεβαίως η Επιτροπή των προγραμμάτων είναι αυτή που αποφασίζει ακριβώς πώς γίνεται η κατανομή στο θέμα της χρηματοδότησης. Αλλά βεβαίως οι προτεραιότητες αναπτύσσονται και αποφασίζονται βάσει των προτεραιοτήτων των κρατών μελών. Υπάρχει ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ και σε καμία περίπτωση δεν αποφασίζονται και δεν διεκπεραιώνονται προγράμματα τα οποία αποτελούν ε, επικαλύψεις σε σχέση με τα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Το θέμα αν τα κονδύλια που διατίθενται για τα αμυντικά και τα εξοπλιστικά προγράμματα, ε, για την έρευνα αυτού του τομέα είναι επαρκή. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω ότι τα κράτη-μέλη εδώ θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της έρευνας. Αυτό που κάνω τώρα το έχω ξαναπεί πολλές φορές αν θέλουμε να παραμείνουμε μπροστά σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Σήμερα υπάρχουν έξι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά εκπροσωπούν το 98% όλης της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα αυτό. Πώς μπορούμε λοιπόν από τη στιγμή που υπάρχουν δεσμεύσει ε, στα προγράμματα PESCO, στα οποία συμμετέχουν 25 κράτη-μέλη. Μα καταλαβαίνετε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι, πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επενδυθεί πολύ περισσότερο στον αμυντικό τομέα, στην έρευνα και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και εννοείται ότι ο προϋπολογισμός αυτός σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί παρά να είναι συμπληρωματικός. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν, να χρηματοδοτούν αυτό τον τομέα. Δεν μπορεί να πούμε ότι αυτό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς ξεχνάμε τη δική μας προσπάθεια. Αν συγκρίνουμε τώρα αυτό που κάνει η Ευρώπη με τρίτες χώρες, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε ότι παλιότερα η Ευρώπη ήταν ένας ακόλουθος αυτών που γινόταν από τους μεγάλους πρωταγωνίστες. Σήμερα δεν ξέρω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται δυνατή προσπάθεια, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στην έρευνα και στην ανάπτυξη και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο συμβατότητας, να υπάρχει δηλαδή διαλειτουργικότητα. Και για πολλούς τομείς της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται ότι θα πρέπει να παραμείνουμε με έναν ρυθμό που δεν θα μας αποκλείσει από τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την άμυνα θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Η Σίλβια θα σας δώσει περισσότερους στοιχεία για τα ποσοστά τους αριθμούς. Μιλήσατε επίσης για την συνοχή μεταξύ των πρωτοβουλειών και των ε, προσπαθειών και πώς μπορούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις. Βεβαίως, συνεχίζουμε τις ε, προσπάθειές μας να παραμείνουμε συνεκτικοί, να έχουμε κοινέ πρωτοβουλίες, όχι μόνο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου και των ε, πρωτοβουλειών που τίθενται από την ΠΕΣΚΟ, αλλά και με τον ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άσκοπες επικαλύψεις. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. 22 από τα μέλη μας είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί λοιπόν να επιλέξουν κάτι τέτοιο. και βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των τριών. Έτσι κι αλλιώς ε, υπάρχει στον σχεδιασμό ο καθοριστικός ρόλος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής που την ίδια ώρα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων των δικών μας και της ΠΕΣΚΟ. Με αυτή λοιπόν την τριπλή ιδιότητα πιστεύω ότι η επιλογή των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων θα γίνει με τρόπο συνεκτικό. Τα κράτη-μέλη, παρόλα αυτά, έχουν αναθέσει στον κύριο Μπορέλ, περί αυτού πρόκειται, την ε, αποστολή να παρουσιάζει κάθε χρόνο μία έκθεση η οποία θα παρουσιάζει τη συνοχή όλης αυτής της πολιτικής. Βεβαίως Υπάρχουν και οι 11 προτεραιότητες της πολιτικής. Υπάρχει το θέμα της δορυφορικής ανάπτυξης προγραμμάτων και βεβαίως το διάστημα, η πλοήγηση. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για το επίπεδο των επενδύσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι να λάβουμε υπόψη μας την αμυντική πτυχή από την αρχή. Να μην ξεκινάμε δηλαδή προγράμματα τα οποία δεν έχουν μια ε, στρατιωτική πτυχή και η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί εκ των υστέρων. για την βιομηχανία, κύριε Πασέσκου, αυτά που είπατε δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εδώ απλά να δηλώσουμε ότι η δήλωση στον αμυντικό τομέα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ε, ένας οποιοδήποτε αμυντικός τομέας με τους ίδιους κανόνες ε, ανταγωνιστικότητας. Αν είχαμε απλώς θέμα ανταγωνιστικότητας της αγοράς, δεν θα ήμασταν ε, σε αυτήν την κατάσταση, διότι καταλαβαίνετε ότι το θέμα ε, εδώ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν ε, τα ίδια δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα όσον αφορά την παραγγελία, την ανάπτυξη την αγορά αυτών των συστημάτων όταν μιλάμε για τον αμυντικό τομέα. Η βιομηχανική στήριξη δηλαδή πρέπει, αν θέλετε, να εξασφαλιστεί αποκλειστικά και μόνο με στήριξη πολιτική. Η οικονομική και πολιτική στήριξη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Χρειάζεται επίσης να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας της εθνικής κυριαρχίας και, και η χρήση αυτών των συστημάτων ε, προϋποθέτει άδεια. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρχει μια τεχνολογική και βιομηχανική βάση η οποία να μπορεί να συνεχίσει να παράγει και μια βιώσιμη αν θέλετε εξοπλιστική βιομηχανία προϋποθέτει συνεργασία. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει με μια ανοιχτή αγορά. Ξέρετε ότι ανοιχτή αγορά στον εξοπλιστικό τομέα, στην αμυντική βιομηχανία δεν μπορεί να υπάρχει, καθότι υπάρχει ένας μόνο πελάτης. Κύριε Λούκας. Well, I, I think uh, in the Νομίζω ότι στη φάση της προετοιμασίας και στους δύο πόλους που ήδη εξετάσαμε, συγκεκριμένα για τη δική σας χώρα, για τη Λιθουανία, η συμμετοχή ήταν πολύ καλή. Και για τη βιομηχανία σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για σας. Και αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον, αλλά όπως σας είπα, πρέπει να αλλάξουμε την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Τι ποσά θα πανώμε για την αμυντική μας βιομηχανία, για τον αμυντικό μας προϋπολογισμό. Τέλος, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, έχω κάποια στοιχεία εδώ. Για το 17, η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου των ε, επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια. Δύο, δύο εκατομμύρια, συγγνώμη, το 17 και ασήμαντο ποσό το 18. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες και βεβαίως ε, με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια όπως εξάλλου συζητήθηκε και αυτά όταν ε, το θέμα ήταν το EIDP και το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Euh, λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Με μεγάλη χαρά ανοίγω αυτήν την ε, ακροαματική διαδικασία για πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτόν εδώ τον Νίκο. Με πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για τα αμυντικά θέματα. Ο κύριος Κιβά δεν μπορούσε να προσέλθει και επομένως έχουμε λόγω σιδηροδρομικού ατυχήματος λέει η Πρόεδρος και επομένως έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες να μας παρουσιάσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα αμυντικά συστήματα. Ο κύριος Ρίπος, ε, υπεύθυνο ερεύνης στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμήνη, ε, υπεύθυνο για θέματα ερεύνη, θα παρουσιάσει τα έργα και τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν. Δεν θέλω βέβαια να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που θα μας πει. Η κυρία Βερμπρούγκεν, ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μελετών, στο ULB, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών θα μας παρουσιάσει τις τρέχουσες ε, συζητήσεις σχετικά με τις συμβάσεις που διέπουν τη χρήση σημαντικών όπλων. Η κυρία Ταντέο στο Ethics Lab θα μας ε, δώσει κάποιες στοιχείες ε, ηθικού προβληματισμού στην χρησιμοποίηση τέτοιων συστημάτων στα αμερικά αισθήματα στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών η ε, τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένα σημαντικό διακύβευμα στρατηγικής φύσεως παγκόσμιο για προγράμματα πολιτικής αλλά και στρατιωτικής χρήσης έχουμε άνευ προηγουμένου εξελίξεις πλέον στην τεχνολογία της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε βαθιές τομές με πολλές καινοτομίες σε διάφορους τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, οι μεταφορές αλλά και η κυβερνασφάλεια και η άμυνα. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να προχωρήσουμε στα θέματα επενδύσεων και ερεύνης το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το μόνο που μπορεί να παράσχει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε το έδαφος που μας χωρίζει από τους πρωτοπόρους γιατί αυτό σχετίζεται με την κυριαρχία μας αλλά και με τον τρόπο ζωής μας και την κοινωνία μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο λοιπόν για χάσιμο στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να λάβουμε σαφείς αποφάσεις και να διαμορφώσουμε ένα απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει τις ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις που θα πρέπει να καλύπτονται. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει το δικό τους πλαίσιο της έρευνας και της χρήσης αυτών των τεχνολογιών, αλλά θα πρέπει να δούμε και λίγο έναν συντονισμό που θα πρέπει να γίνει μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων. Από το 2014 έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνείδηση κοινή σχετικά με το θέμα αυτό, με την, Ευρωπαϊκή, με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τεχνητή νοημοσύνη για την Ευρώπη, αξιόπιστη χρήση τη τεχνολογίας αυτής. Διερωτάται λοιπόν κανείς γιατί τόσο καιρό έχουμε μείνει απλώς στο στάδιο των παρατηρήσεων της θεωρητικής σκέψης, εξέτασης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει, δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε να χάσουμε περισσότερο χρόνο σχετικά με αυτό. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί στα 100 πρώτες μέρες της εντολής της να παρουσιάσει ένα σχετικό πλαίσιο σχετικά με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτής που μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς ε, οργάνωση, συλλογής ε, και επεξεργασίας δεδομένων ολόκληρος ο πλανήτης επενδύει μαζικά ε, στις τεχνολογίες αυτές δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει στο περιθώριο και γι' αυτό παρατηρούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τα αισθήματα ε, τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των αμυντικών ζητημάτων. Έχουμε και το EDIDP, ε, το πρόγραμμα της στρατηγικής αυτονομίας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διατηρήσουμε την αυτονομία μας μακροπρόθεσμα. Ελπίζουμε ότι οι τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιθετικά στο πλαίσιο αυτό να είναι και μεταξύ των επιλεξίμων δράσεων υπό το μελλοντικό Ταμείο Αμήνης. Έχουμε εδώ ένα δυναμικό για να βελτιώσουμε τη δυνατότητα παρέμβασής μας ταχαίως και αποτελεσματικός ιδιαίτερα στα πλαίσια στρατιωτικών αλλά και πολιτικών αποστολών όπου αντιμετωπίζουμε πολλές και διάφορες προκλήσεις. Οι ηθικές πτυχές διαστάσεις των αυτόνομων συστήματων στόχευσης των επιθετικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη ε, προκαλούν έντονη ανησυχία. Υπάρχει μία αναζήτηση σχετική με το επίδο της ευθύνης του ανθρώπινου χρήστη, του ελεγκτή δηλαδή, ε, όλα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν σε ένα πλαίσιο ταχεία λήψη απόφασης. Επίσης, υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για την ε, χρησιμοποίηση φωνικών όπλων σχετικά με την ανάπτυξη οποιοδήποτε αυτόνομου συστήματος επιθετικού που χρησιμοποιεί φωνικά όπλα στόχευση και ότι αυτό θα έπρεπε να είναι υπό ανθρώπινο έλεγχο. Και αυτά τα συστήματα έχουν αποκλειστεί από τα επιλέξιμα όμως ε, έργα υπό το μελλοντικό ταμείο. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συντονισμένη προσπάθεια να συνδιαμορφώσει μια προσέγγιση σχετικά με τον περιορισμό κάποιων οπλικών συστημάτων. Προτού δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, να επαναλάβω ότι είναι άμεση η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η όθηση για την εκκίνηση διεθνών διαπραγματεύσεων στο θέμα αυτό, ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Επιθυμούμε μια τεχνητή νοημοσύνη ευρωπαϊκή θα την έλεγα, ισχυρή αλλά και ελεγχόμενη από τον άνθρωπο και τις ηθικές του αρχές που να μπορεί να ελέγχεται σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, ξεκινώντας από τον κύριο Ρυπός. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω για το ζήτημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υπόθηκε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί νέο θέμα όσον αφορά τις πιθανές τεχνολογίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για αμυντικές εφαρμογές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η διαχείριση των πολύ μεγάλων δεδομένων, των σχετικών λογισμικών προγραμμάτων στον τομέα της πληροφορικής. Έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο με αποτέλεσμα τεχνητή νομοσύνη να γίνει πλέον πραγματικότητα. Η νέα αυτή πραγματικότητα συνδυάζεται με κάποιες ε, εμπορικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των πρωτοβουλειών αυτών στον αμυντικό τομέα και πολλά παραδείγματα μπορείτε να δείτε ακόμα και στον τύπο. Τώρα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά στον τομέα της άμυνας, εδώ πρέπει να, την, να τονίσουμε ότι ε, οι σχετικές αποφάσεις που θα ληφθούν στον τομέα της τεχνολογίας θα αλλάξουν εντελώς το πεδίο το τοπίο της άμυνας όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Θα οδηγήσουν σε νέες επιδόσεις, νέες ανάγκες, νέες δεξιότητες, νέο τεχνικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και σε νέα αμυντικά δόγματα και νέες αμυντικές διαδικασίες. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι καθοριστική σημασία και να αλλάξει εντελώ το τοπίο, μπορεί να οδηγήσει σε νέα διεξαγωγή των συγκρούσεων, σε διαφορετική συμπεριφορά των ενόπλων δυνάμεων και στη διαφορετική αντιμετώπιση του άμαχου πληθυσμού. Για παράδειγμα, ενδεχομένως η χρησιμοποίηση της τεχνικής, ε, τεχνητής νοημοσύνης να οδηγήσει σε λιγότερες ε, παράπλευρες απώλειες στο πλαίσιο μιας μάχης, καθώς ε, η χρησιμοποίηση οπλικών συστημάτων θα είναι πιο μικρή και πιο στοχευμένη. Μπορούν να οδηγηθούμε επίσης σε χαμηλότερες δαπάνες, σε χαμηλότερο κόστος. Ωστόσο, η έγκριση αυτή των νέων, τεχνητών των νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε νέες αδυναμίες και νέα τροτά σημεία. Μπορούμε να έχουμε μια χειραγώγηση των πληροφοριών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για καμπάνιες παραπληροφόρησης, χειραγώγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά μπορεί ψυχολογικά να πειράσουν πάρα πολύ μια στρατιωτική επιχείρηση. Πρέπει επίσης να πούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να γίνουν επιθέσεις με τρόπο πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο επιζήμιο. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το ζήτημα της προστασίας και της ασφάλειας. Λοιπόν, πρέπει να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο πιο αξιόπιστο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο εμπιστοσύνη, πάρα πολύ είναι ιδιαίτερα διστακτική απέναντι στη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη και στα αποτελέσματα που μπορεί αυτή να φέρει. Τώρα, ποιο μπορεί να είναι ο αντίκτυπο όσον αφορά το τομέα τη άμυνα. Μία από τι βασικέ υποσχέσει που μα δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι στον τομέα της άμυνας η εφαρμογή της μπορεί να είναι τόσο ευρεία που μπορεί να έχει τελικά πολλές διαφορετικές επιπτώσεις. Στο στρατιωτικό λοιπόν πεδίο η τεχνητή νομοσύνη μπορεί να βρει εφαρμογή παντού, στην εναέρια, χερσαία, θαλάσσια άμυνα, ακόμα και στην κυβερνοάμυνα και σε παντού, παντός είδους συγκρούσεις, στρατηγικές, τακτικές και το καθεξής και μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί πλέον στο τμήμα μιας ασύγχρονης σύγκρουσης. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις και σε συγκεκριμένες στρατιωτικές αποστολές, οι οποίες μπορεί πλέον να διεξάγονται πολύ πιο γρήγορα σε ένα πολύ πιο πολύπλοκο περιβάλλον. Θα υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα, και θα μπορούμε να ανταποκριθούμε πολύ πιο γρήγορα σε πολύ, πολύ διαφορετικές ε, αποστολές και επιχειρήσεις. Επίσης, ε, μπορούμε πλέον να διεξάγουμε πολύ πιο γρήγορα επιχειρήσεις, οι οποίες αν διεξάγονταν μόνο από τον άνθρωπο, θα θεωρούνταν ιδιαίτερα χρονοβόρες ή θα δοκίμαζαν πάρα πολύ την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Μπορούμε επίσης ε, να διεξάγουμε πολύ πιο γρήγορα επιχειρήσει οι οποίε θεωρούνται πολύ πιο επικίνδυνε ή που λογικά θα πετούσαν πολύ περισσότερου στρατιώτε. Η που θα πετουσαν πολυ χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε νέες εφαρμογές όσον αφορά τη χρήση υπολογιστικών γλωσσών, ρομποτικής και άντλησης δεδομένων. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση, την αναγνώριση, την ανάλυση πληροφοριών, την εκπαίδευση, την στρατιωτική κατάρτιση και το καθεξής. Βέβαια, προκειμένου να καταλάβουμε πραγματικά τις επιπτώσεις μπορεί να έχει τεχνητή νοημοσύνη στη διεξαγωγή πολέμων, θα πρέπει να δούμε πραγματικά πώς μπορεί αυτή να βελτιστοποιήσει τις συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται και πώς αυτές έπειτα θα αξιολογηθούν από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, διαφαίνονται διάφορες ευκαιρίες ε, από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ένας πρώτος τομέας εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι η ε, αναγνώριση, η συλλογή πληροφοριών, η καλύτερη αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίε θα μπορούσαν να καταστούν πολύ πιο συγκεκριμένε. Θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να μπορούμε να αντιδρούμε πολύ πιο γρήγορα και να λαμβάνουμε πολύ πιο γρήγορα αποφάσει. Θα μειωθεί κατά αυτόν τον τρόπο φόρτο εργασία, καθώ επίση και οι ανάγκε κατάρτιση όσον αφορά του χειριστέ των ανιχνευτήρων. Επίση, μπορούμε να αυξήσουμε μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη την επιχειρησιακή μα ετοιμότητα και να κάνουμε έναν εξορθολογισμό της διοικητική μέρημνα και τη συντήρηση και κατά αυτόν τον τρόπο να προβούμε και σε εξοικονόμηση πόρων. Επενδύοντας στη τεχνητή νοημοσύνη θα μειωθούν οι επιχειρησιακέ δαπάνε και θα προστατεύσουμε καλύτερα τον στρατό μα αλλά και τον άμαχο πληθυσμό, για παράδειγμα βελτιώνοντας την ακρίβεια του στόχου. Τώρα, όσον αφορά τις προκλήσεις, Τέσσερις βασικές προκλήσεις έχουμε εντοπίσει. Πρώτον, διαχείριση των δεδομένων, διαχείριση των big data και επιμερισμός των δεδομένων αυτών. Στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, στην, στο machine learning χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο αριθμό αντιπροσωπευτικών δεδομένων αλλά ξέρετε ότι είναι πραγματική πρόκληση το να διαχειρίζεται κανείς από κοινού τέτοια δεδομένα στον τομέα της άμυνας, σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας. Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα εμπιστευτικά, ευαίσθητα, πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα σε μεγάλο αριθμό και δεν υπάρχει απαραίτητη ευελιξία πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Τα ζητήματα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιληθούν προτού εφαρμόσουμε ένα κοινό σύστημα, μια κοινή διαδικασία συλλογής δεδομένων. Έπειτα πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριμένες κοινέ διαδικασίες σε διεθνές επίπεδο για τη συλλογή των δεδομένων αυτών. και αυτό με τη σειρά του θέτει κάποιες προκλήσεις, αν μιλάμε για συλλεγή δεδομένων ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες στον τομέα της άμυνας, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση δεδομένων για τη διοικητική μέρημνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή, η οποία έχει διάφορες τεχνικές, τεχνολογικές πτυχές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές νομοθεσίες στον εμπορικό τομέα που εμποδίζουν τελικά την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά από τη μία χώρα στην άλλη. Η χρήση λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης καλείται πραγματικά να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή και να προωθήσει τελικά μια διεθνική συνεργασία όσον αφορά την άντληση και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών. Άρα χρειαζόμαστε μια πολύ πιο σύγχρονη αρχιτεκτονική στην άντληση και τη διαχείριση των δεδομένων αυτών. Θα πρέπει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα αυτά σε όλο τον κύκλο ζωής τους και η οργάνωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στον τομέα της άμυνας είναι αρκετά κατακαιρματισμένη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές ομάδες δεδομένων και διαφορετικά μεγέθη δεδομένων. Πολλές φορές τα δεδομένα που έχουμε δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να οργανώνουμε τα δεδομένα αυτά, πώς θα μπορούμε να φιλτράρουμε αυτά τα δεδομένα, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά, πώς μπορούμε να τους επιφέρουμε προσαρμογές και αλλαγές και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλη την αλυσίδα διαχείριση δεδομένων πανευρωπαϊκά και αυτό από μόνο το αποτελεί πολύ μεγάλη πρόκληση. Όσον αφορά τώρα την πιστοποίηση των δεδομένων αυτών, Πάλι εδώ πέρα θα χρειαζόμαστε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα μπορούν να πιστοποιούν τα δεδομένα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει μια κατάρτιση των μηχανών αυτών και να μπορούμε να διασφαλίσουμε σε τεχνικό επίπεδο ότι θα υπάρχει μια ομοιόμορφη λειτουργία των μηχανών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και μια συγκεκριμένη πιστοποίηση για τις μηχανές αυτές που θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την άντληση και την επεξεργασία των δεδομένων. Και ας μην παραβλέπουμε βέβαια ότι μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι χειριστές, οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν και αυτοί με τη σειρά τους πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα και πολλές διαφορετικές πιστοποίησεις από τη μία χώρα στην άλλη και εν γέννη. Οι διαφορετικοί αυτοί κανονισμοί και οι διαφορετικές αυτές πολιτικές υστερούν σε σχέση με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών αυτών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε με τα διάφορα workshops τα οποία διοργανώνουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινή λειτουργική κατανόηση για τα συστήματα αυτά και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους χρήστες που θα κληθούν να επεξεργαστούν αυτά τα συστήματα. Όσον αφορά τώρα την καινοτομία και την ελκυστικότητα, εδώ θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι βασικέ εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη ξεκινήσει από το μη στρατιωτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τις εφαρμογές αυτές τεχνητές νοημοσύνης στις ανάγκες του τομέα της άμυνας. αυτό το εγχείρημα όμως ε, ενδεχομένως να περιπλακεί αν δεν έχουμε τις απαραίτητες ε, δεξιότητες. Θα πρέπει λοιπόν ε, στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τις πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν στο μη στρατιωτικό τομέα, προκειμένου να πτύξουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα είναι ανοιχτά από τεχνολογικής πλευράς και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο τομέα της άμυνας. Να φέρουμε εδώ πέρα στο ανοιχτό λογισμικό ή σε αλγόριθμους οι οποίοι εκπονήθηκαν για το μη στρατιωτικό τομέα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και στον τομέα της άμυνας. Και υπάρχουν βέβαια και οι πτυχές που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια, οι οποίες ε, και αυτές σχετίζονται άμεσα με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η αμυντική κοινότητα επί του παρόντος προσπαθεί να δει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τροποποιήσει βασικές λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε προτού η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιείται εν γέννη. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να ενσωματωθεί στον τρόπο που λειτουργεί ο τομέας της άμυνας και στον τομέα που εξελίσσεται από την ad hoc χρήση της μέχρι την ενσωμάτωσή της σε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες προβληματικές πτυχές, όπως για παράδειγμα διαδικασίες απόκτησης αγοράς. Ξέρετε ότι με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τα συστήματα αγοράς αμυντικού εξοπλισμού. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούν τα αμυντικά δόγματα και οι επιχειρησιακές αμυντικές διαδικασίες οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, καθώς επίσης και το νομικό πλαίσιο και το δοντολογικό πλαίσιο. Όλα αυτά όμω θα πρέπει να γίνουν αν πραγματικά θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να ενσωματωθεί στα προγράμματα τα αμυντικά τι επόμενε δεκαετίε. Προτού ολοκληρώσω, να αναφερθώ, να αναφερθώ λίγο στις, αμυντικ... στις νομικές και διοντολογικές πτυχές, ζητήματα τα οποία θα καλύψουν ε, εις βάθος οι επόμενοι ομιλητές η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα φωνικά αυτόνομα οπλικά συστήματα είναι σαφής. Η χρησιμοποίηση βίας θα πρέπει πάντα να διέπεται από το διεθνές δίκαιο και θα πρέπει τα φωνικά αυτά αυτόνομα οπλικά συστήματα να υπάγονται πάντα στην ανθρώπινη ευθύνη. Όπως ε, ε, είπαν ε, Άλλωστε και η αρμόδη σε μια άλλη ακρόση που οργανώθηκε τον Σεπτέμβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάλι από το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους που αναφέρεται συγκεκριμένα στα φωνικά αυτόνομα οπλικά συστήματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θα κάνουμε με τις επαναστατικές αυτές νέες τεχνολογίες και πώς μπορεί να εμπλεκεί όμως και η κοινωνία των πολιτών στις αποφάσεις που θα ληφθούν και όσον αφορά τις αξίες που θα πρέπει να διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό στο εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, η ανάπτυξη κάποιων τοπικών οικοσυστημάτων δεξιοτήτων είναι εξή πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που θα προκύψουν στον αμυντικό τομέα από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές, είτε πρόκειται για την έρευνα, είτε πρόκειται για την συμμετοχή της βιομηχανίας, είτε πρόκειται για την κάλυψη των αμυντικών απαιτήσεων και θέλουμε να προωθήσουμε εμεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα ένα κοινό αφήγημα όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τη τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα τη άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκπονούμε επίση ένα έγγραφο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, όσον αφορά τον, τους όρους που χρησιμοποιούμε στη τεχνική νοημοσύνη, τις βασικές αρχές Τη ε, τεχνητή νοημοσύνης προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στις γενικότερες προσπάθειες ενημέρωσης που, που γίνονται όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της τεχνητή νοημοσύνης στην αμυντική έρευνα. Όπως σας είπα, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη πραγματικότητα από το 2016 είχαμε περίπου 30 προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία προωθήθηκαν από τις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και 12 προγράμματα θεωρούνται ad hoc, στα οποία συμμετέχουν εκ περιτροπής τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό προγραμμάτων που χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Βάσει των διαφορετικών αυτών δραστηριοτήτων και των μελετών που έχουν γίνει από τα κράτη-μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, προσπαθούμε να αποτιμήσουμε τις ευρωπαϊκές αμυντικές στρατηγικές και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα προσπαθεί να εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση για τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα. Στι αρχέ του 2020 θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του σχεδίου αυτού δράσης να σας δώσω κάποια, προγράμματα από, κάποια παραδείγματα με συγχωρείτε, από τα εργαστήρια, εργαστήρια αυτά που χρησιμοποιούμε μια προσωμείωση τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιούμε την κάνουμε μάλλον έρευνες όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην χρήση ραντάρ. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα συμβάλλει στην αμυντική καινοτομία και θα έχουμε και ένα ακόμα εργαστήριο όσον αφορά τις γλώσσες στον τομέα της τεχνολογίας. Ολοκληρώνω την παρουσίασή μου αυτή τονίζοντας ότι ε, η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της άμυνας μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά νέες ευκαιρίες, δημιουργεί νέους ε, ρυθμούς διεξαγωγής ε, των συγκρούσεων και είναι όλο και πιο παρούσα στον αμυντικό τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι τεχνολογικές αυτές αποφάσεις επηρεάζουν όλες τις διαφορετικές πτυχές του αμυντικού τομέα και είναι πάρα πολύ σημαντικό η τεχνητή αυτή νοημοσύνη να ενσωματωθεί σε όλες τις αμυντικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις δεξιότητες, ε, την χρήση της πληροφορικής στον τομέα των ε, αμυντικών συμβάσεων και το καθεξής. Πολλές διαφορετικές μπορεί να είναι οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στους τομείς αυτούς και ο επότερο στόχος είναι να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να χρησιμοποιούν όλο και πιο αποτελεσματικά στις ένοπλες δυνάμεις τους στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βέρμπρουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι σήμερα εδώ. λέγαμε Μαρία Κεφερμπράχα και εργάζομαι στην, ε, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο εδώ στις Βρυξέλλες. Κάνω έρευνα σε θέματα στρατιωτικής καινοτομίας και ρύθμισης της ε, τεχνητής νοημοθήνης. Θα σας μιλήσω για τα συστήματα, τα λεγόμενα αυτόνομα φωνικά οπλικά συστήματα, τα περίφημα LOS και θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποια απορίσματα με σκοπό να φτάσουμε σε μια ομοφωνία και συστάσεις για το Κοινοβούλιο. Βέβαια δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το θέμα της αυτονομίας. Κατά πόσο είναι αυτόνομα και περί αυτού πρόκειται. Δεν αναφερόμαστε σε καμία περίπτωση για την αντικατάσταση των ανθρώπινων όντων από ρομπότ ε, της Συζητούμε όμως ε, για μία ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την επιλογή των στόχων. Και βεβαίως εδώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλά επίπεδα. For instance, ε, Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να εντοπιστούν κάποια ειδικά τεθωρακισμένα, εντοπίζονται βάσει του ε, σχεδίου τους, ε, του σχήματός τους. Ε, το ίδιο ακριβώς γίνεται και με σκάφη βάση της <clears throat> ταυτότητάς τους, του σχήματός τους. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο μπορεί ένας στρατιώτης, ο οποίος να αντικατασταθεί ενδεχομένω από την τεχνική νοημοσύνη, να εντοπίσει αυτούς του στόχου, Γιατί λοιπόν εδώ αναφερόμαστε για κάποιες προβληματικές πτυχές αυτής της αντικατάστασης. Υπάρχουν χώρες οι οποίες συμφωνούν ότι δεν θα ήταν σωστό να δημιουργηθούν πλήρως αυτόνομα συστήματα τα οποία θα εντοπίζουν μόνοι τους τους στόχους και θα τους ε, εξαλείφουν χωρίς καμία παρέμβαση των ανθρώπων. Ποιο είναι ο ανθρώπινος έλεγχος που είναι απαραίτητο, ποια είναι τα στοιχεία αυτά της δραστηριότητα αυτής τα οποία θα πρέπει να γίνονται αυτόνομα. Το ερώτημα είναι αν αναφερόμαστε μόνο σε επιθετικά συστήματα ή αν αναφερόμαστε και στα αμυντικά. Και το θέμα είναι ότι παραδείγματο χάνει συστήματα αεράμινα ε, με κάποια αυτονομία χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Ποιε είναι οι αυτοματοποιημένε πτυχέ αυτών των συστημάτων, ποιε είναι οι αυτόματε πτυχέ του, σε πιο προηγμένα συστήματα, πιο αυτόνομα συστήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο, διότι το βαθμός της αυτονομίας είναι αλληλένδετος. Υπάρχει βεβαίως εδώ και μια σχετική αυτονομία των συστημάτων, αναφερόμενο σε κάποια φουτουριστικά συστήματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Θα ήθελα να αναφερθώ στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, σε κάποιους πυράβλους, αλλά συστήματα τα οποία ουσιαστικά προτείνουν στον άνθρωπο τον εντοπισμό κάποιων στόχων. Η απάντηση της μηχανής, η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πολλές φορές να συμπληρώσει την κρίση των ανθρώπων. Το θέμα είναι αν είναι νόμιμο, αν είναι επιθυμητό και πάντα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι φοβούνται υπερβολικά τα μηχανήματα, τις μηχανές. Αντίθετα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος πολλές φορές είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με τα αυτοματοποιημένα συστήματα που βασίζονται στην τεχνική νομοσύνη. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο θέλει ο άνθρωπος να χάσει τον έλεγχο εδώ όσον αφορά τον εντοπισμό και την εξάλληψη των στόχων. Επίσης, ένας κανονισμός για τη ρύθμιση αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό βήμα. Η αυτονομία λοιπόν είναι προβληματική. Μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχουν θέματα ηθικά, δεοντολογικά και θέματα ασφάλειας. Το βασικό νομικό θέμα όμως είναι αν η αυτόνομη χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να αντιτεθεί ή να συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Υπάρχουν σαφώς προδιαγραφές και απαιτήσεις των οπλικών συστημάτων και κάποιες νομικές δεσμεύσεις, οι οποίες βεβαίως ε, θα πρέπει να, να κάνουν τη διάκριση μεταξύ αμάχων και στρατιωτών. Ποιος μπορεί να πάρει την απόφαση και βάσει ποιον προδιαγραφών και συντελεστών Επίσης, πώς μπορεί να πάρει την απόφαση κάποιος πριν την εκτέλεση μιας απόφασης. Η στόχη, η νομική ανάλυση αυτών ο βαθμός αυτονομίας και πώς και πότε μπορεί να παρέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας. Βεβαίως εδώ δεν απαιτείται από τους στρατιωτικούς να παρέμβουν μετά την ολοκλήρωση ενός συστήματος. Οι συνθήκες βεβαίως μπορεί να αλλάξουν μετά το ξεκίνημα μιας επιχείρησης και εδώ βλέπουμε ότι ο καθορισμός κάποιων στόχων, κάποιων συγκεκριμένων στόχων, μπορεί πολλές φορές ε, να εμπλέκεται και με την παρουσία άμαχου πληθυσμού. Υπάρχουν λοιπόν πορύπλοκες αποφάσεις, υπάρχει η αλυσίδα της απόφασης, η λογοδοσία κατά τη διάρκεια και στο τέλος μιας επιχείρησης. Το θέμα της λογοδοσίας, από τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει ένας συγκεκριμένος βαθμός αυτονομίας αυτών των συστημάτων, αλλά και ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς και όλα τα προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζει μία απόφαση βάσει τεχνικής νοημοσύνης. Ποιος θα είναι υπεύθυνο, Υπάρχει θέμα λογοδοσίας και συμβατότητας και βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα αντίθετο επιχείρημα όσον αφορά την ήδη υπάρχουσα χρήση αυτόματων συστημάτων βάσει των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τα δεοντολογικά και ηθικά αυτά επιχειρήματα μας οδηγούν από τη μία στην χρήση αυτών των αυτόματων φωνικών συστημάτων με την έννοια ότι δεν έχουν συναισθήματα και ότι θα μπορέσουν σίγουρα να είναι πιο αντικειμενική η χρήση τους να μην καθοδηγούνται από τα συναισθήματά τους και να μην ασκήσουν σεξουαλική βία. Το θέμα όμως των ε, αντίθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας ε, επιχείρησης και η χρήση αυτών των αυτόματων ε, φωνικών συστημάτων είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την παρέμβαση και τον έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα, με περισσότερη ε, παρουσίαση και έλεγχο των νομικών κειμένων που διέπουν αυτή τη χρήση. Τέλος, ακριβώς ε, επειδή υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ των ε, ηθικών πτυχών αυτής της χρήσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα διάφορα επίπεδα ε, διοίκησης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα νομικά κείμενα να μας προστατεύουν κατά τέτοιων αποτρόπαιων χρήσεων και εγκλημάτων. Υπάρχουν πολλές πτυχές όπως το θέμα της, ε, του επίπεδου επέμβασης και παρέμβασης αυτών των συστημάτων. Η αυτονομία αυτών των συστημάτων θα δημιουργήσει περισσότερα θύματα ή θα μειώσει την ε, παρουσία ανθρώπων στις επιχειρήσεις. Η κλιμάκωση των ε, επιχειρήσεων, η παρέμβαση των ε, ανθρώπων που πολλές φορές δεν δικαιολογείται από το μέγεθος και το βαθμό της απειλής, ιδιαίτερα όταν παραδείγματος χάνει αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο αυτά τα αυτόνομα συστήματα. Δεν είναι εύκολο να δει κανείς πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία αυτών των συστημάτων. Τέλον, είναι σημαντικό να υπάρξει νομική πλαισίωση αυτών των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαφορετικά επιχειρήματα. Αυτό είναι κάτι διαπιστώνουμε ότι η δημόσια, η κοινή γνώμη δεν έχει ακόμα δεχθεί αυτά τα ηθικά επιχειρήματα. Ήδη από το 2014 συζητήθηκε το θέμα αυτό στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για τα συμβατικά και τα νέα οπλικά συστήματα και υπάρχουν πολλές διαφορετικές προτάσεις. Έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις οι συζητήσεις συνεχίζονται ακόμα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η ρύθμιση και οι κανονισμοί που θα οδηγούσαν σε μία πλήρη απαγόρευση αυτών των αυτόμανων συστημάτων ή η επιλογή μίας ανθρώπινης παρέμβασης, έναν ανθρώπινου ελέγχο. Μέχρι τώρα υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά την ανθρώπινη παρέμβαση, τον ανθρώπινο έλεγχο. Μία άλλη εναλλακτική θα ήταν μια πολιτική δήλωση για την μη χρήση αυτών των οπλικών συστημάτων, η οποία όμως δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων αυτών, η χρήση νέων οπλικών συστημάτων αυτόνομων, καθώς και η περιορισμένη τους δυνατότητα ανάπτυξης. Βλέπουμε όμως ότι Συζητήσει συνεχίζονται στη Γενέβη στα πλαίσια των Ηνωμένων Αθήνων και πριν από ορισμένε εβδομάδε. Μήπω μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά. Η έλλειψη συμφωνίας και ομοφωνίας ουσιαστικά βασίζεται εδώ σε πάρα πολλούς παράγοντες. Υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τι ακριβώς ε, είναι το θέμα της ε, νομικής δέσμευσης και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες και ορισμοί όσον αφορά την αυτονομία αυτών των συστημάτων. Και παρόλο που πολλές φορές ε, μπορεί οι εμπειρογνώμονες να συμφωνήσουν, στην πράξη υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Παραδείγματο χάρη, πότε είναι μια λειτουργία αυτόνομη όταν ένα σύστημα είναι πλέον ανεξέλεγκτο και πώς η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να έχει κάποιο το αποτέλεσμα βλέπετε ότι αυτός ο ορισμός είναι κενός και δεν υπάρχει απολύτως καμία συμφωνία μεταξύ των ειδικών. Οι περισσότερες χώρες δεν έχουν σαφή πολιτική, διότι ακριβώς δεν ξέρουν πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία στο μέλλον και επειδή θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει ακόμα η εσωτερική συζήτηση για το ποιο θα πρέπει να είναι το μέλλον που θα επιλέξει η κάθε χώρα. Η πλήρης απαγόρευση, ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν επενδύσει πολύ στην έρευνα και ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να αποφασιστεί. Επίσης, όταν παραμένουν ανοιχτές οι επιλογές για ανάπτυξη των οπλικών αυτών συστημάτων από άλλες χώρες. Τα υπάρχοντα οπλικά συστήματα, όπως αυτά τα οποία προηγουμένως αναφέραμε, το σύστημα Goalkeeper, το οποίο δύσκολα μπορεί να επαληθευτεί κατά πόσο συνεχίζει η ανάπτυξη αυτών των λογισμικών. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν αυτές ε, οι συγκεκριμένες αναπτύξεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εκτός του στρατιωτικού τομέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε προς ποια κατεύθυνση θα ληφθεί η απόφαση από τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στη Γενέβη. Και βεβαίως, στα πλαίσια των ΗΠΑ, το CCW συνεχίζει την συζήτηση με τη συμμετοχή πολλών κρατών μελών. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει προς ποια κατεύθυνση θα συνεχίσει η διαπραγμάτευση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα μπορούσε να κάνει για να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτές τις ε, συζητήσεις. Οι περισσότερες συζητήσεις παρόλα αυτά παραμένουν αρκετά γενικές. Διάφορα σενάρια για διαφορετικά συστήματα και αυτόνομες λειτουργίες. Ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα και γιατί τα νέα αυτά οπλικά συστήματα διαφέρουν αποτελεσματικά από τα υπάρχοντα. Βεβαίως υπάρχει σύγχυση και δεν υπάρχει συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεχίσει τη συζήτηση έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές και οι κυβερνήσεις να συμμετάσχουν περισσότερο και να αυξηθεί η ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Τέλος, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παράδειγμα το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποκλείσει την οποιαδήποτε χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου για τέτοια αυτόνομα οπλικά συστήματα. Δεν νομίζω όμως ότι κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η οποιαδήποτε συμμετοχή και η οποιαδήποτε επιτήρηση και έλεγχος από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπέρος, πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσει για το πώς αναπτύσσονται αυτά τα νέα οπλικά συστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στην οποιαδήποτε ερώτηση. Merci, Ευχαριστούμε κυρία Ταντέο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μπορώ να είμαι μαζί σας. Ε, σήμερα η περιγραφή μου λέει ότι είμαι φιλόσοφος, επομένως ίσως να έχετε μια έντονη τάση να διαφύγετε από την αίθουσα, ελπίζω να μην σας κουράσω. Θα ξεκινήσω με έναν ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορούμε να την κατηγοριοποιήσουμε, κυρίως μέσω της δομής της αρχιεκτονικής της, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρσι, την ορίσαμε ως τον αυξανόμενο πόρο της αυτοδιδασκόμενης οντότητας που μπορεί να εκτελεί καθήκοντα που διαφορετικά η ανθρώπινη νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης επιτυχώς να εκτελέσει. Η φύση λοιπόν αυτής της ευφυΐας, αυτής της οντότητας εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τα ανθρώπινα συναισθήματα, τις ανθρώπινες τάσεις, την ανθρώπινη ευφυΐα. Μιλούμε για την εκτέλεση δράσεων, μιλούμε για την μίμηση της ανθρώπινης δράσης. Επομένω, ε, όλα αυτά τα παραδείγματα, τα οπλικά συστήματα, οι σούπερ ευφυΐες, όλα αυτά είναι, ε, ε, είναι χρησιμοποιούνται περισσότερο στην ε, περιοχή του κινηματογράφου και του μυθιστορήματος ε, και όχι με την πραγματικότητα. Εδώ ασχολούμαστε με τη φύση λοιπόν της διαδραστικής αυτής οντότητας που διδάσκει τον εαυτό της. Αυτό είναι η πηγή όλων των ηθικών προβλημάτων που εξετάζουμε όταν μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις. Δεν θα ασχοληθώ με όλες από αυτές. καταρχάς επιτρέπουν το ανθρώπινο έγκλημα, περιορίζουν τον ανθρώπινο έλεγχο, υποσκάπτουν τα, τις ανθρώπινες δεξιότητες και επιτρέπουν και μια κλιμάκωση αντιπαράθεσης. Αυτά τα προβλήματα είναι πολύ σημαντικά όταν μιλούμε για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Καταρχάς έχουμε το θέμα του ελέγχου. Τα περισσότερα συστήματα AI, ιδιαίτερα τα πιο εξελιγμένα παραμένουν κλειστά κουτιά. Μπορούμε να δώσουμε ένα input, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το output. Ούτε μπορούμε να το εξηγήσουμε αναγκαστικά. Και μιλούμε από την ιατρική διάγνωση μέχρι τα αμυντικά συστήματα, μέχρι τους, ε, ε, τις κρίσιμες υποδομές. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε ασφαλή πρόγνωση του αποτελέσματος του πώς θα δράσει. Θα θυμάστε τον Blade Runner στο σινεμά. Δεν είναι... Αυτό μας θυμίζει απλώς, είναι ένα άλλο κίνδυνο. Ότι έχουμε μια ανθρωπομορφική τεχνολογία υπό μια έννοια. Αλλά θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι παραμένουν υπεύθυνοι και για τις επιτυχίες και για τις αποτυχίες των συστημάτων αυτών. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διατήρηση των δεξιοτήτων μας. Μιλούμε για την αγορά εργασίας, μιλούμε για τα επαγγέλματα, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη για την κυβερνασφάλεια π.χ. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι αναλυτές, οι εμπειρογνώμονες μπορούν να ταυτοποιήσουν μια επίθεση μπορούν να αντιδράσουν, να την αντιμετωπίσουν. Πρέπει να μπορούμε να αναθέτουμε καθήκοντα. Ιδάλλως δεν θα γνωρίζουμε πότε η τεχνητή νοημοσύνη ή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υφίσταται επίθεση και λειτουργεί ή όχι. Αυτό είναι ένα πλαίσιο λοιπόν εισαγωγής στα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία. Εδώ έχουμε ένα, μια δυναμική χαρτογράφηση, απεικόνηση που ο οργανισμός ΝΟΡΣ ε, έχει στην ιστοσελίδα του και δείχνει άνω των 4.000 επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα. Θα έλεγε κανεί, αυτά ήταν το 14, σήμερα θα έχει βελτιωθεί σίγουρα η κατάσταση. Όχι. Το Παγκόσμιο Φόρουμ μας λέει ότι το 2019 η επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ήταν στις πέντε μεγαλύτερες πηγές σημαντικών παγκοσμίων κινδύνων. Γεμάλτο αναφέρει ότι στο πρώτο εξάμεινο 18 ε, έγινε επίθεση σε 4,5 δισεκατομμύρια αρχεία που είναι το διπλάσιο ολόκληρου του έτους 2017. Η Microsoft δείχνει ότι 60% των επιθέσεων του 18 διήρκεσαν κάτω από μία ώρα και χρησιμοποίησαν νέε μορφές επιθετικού λογισμικού malware τέλο πάντων. Ποια είναι η δυναμική που περιγράφει όλα αυτά. Εδώ μας βοηθάει λίγο η φιλοσοφία. Όταν μιλούμε για μη κινητικές κυβερνητικές επιθέσεις, δηλαδή όχι αυτές που φωνεύουν κανονικά, αλλά μένουν εικονικές, είναι εύκολο να τις ξεκινήσει κανείς παραμένοντας στην ανωνυμία και με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό τεχνικώς το αποκαλούμε περιβάλλον σταθερά επιθετικό. Πάντα προσπαθούμε να επιτεθούμε. Γίνονται απόπειρες διαρκής αναζήτηση μέχρι να βρούμε ένα κενό στο σύστημα άμυνας. Και εδώ μιλούμε για τον εξοπλισμό του κυβερνοχώρου. Και ε, συνθέτεται ένας κύκλος, ένας φαύλος κύκλος, εάν προσθέσουμε και τους ε, κυβερνητικούς ή κρατικούς φορείς, τότε αυτοί οι φαύλοι κύκλοι γίνονται ακόμα ταχύτεροι. Η τεχνητή νοημοσύνη εδώ έχει σημαντικότερο ρόλο να διαδραματίσει ένα τέτοιο σενάριο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλή στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αντεπίθεση. Αυτό το μάθαμε το 2016 με, διάφορες, με διάφορα κρούσματα συγκεκριμένα με, με το πολεμικό παιχνίδι Capture the Flag επίσης για παράδειγμα ώστε να ταυτοποιούνται τα κενά οι αδυναμίες του ε, συστήματος που ε, αμήνεται ή του συστήματος που επιθυμούμε να επιτεθούμε εναντίον του. Και όλα αυτά δεν αφορούν σε κάποιο απότερο μέλλον. Όταν μιλούμε για, την, για το πόσο ισχυρά είναι τα συστήματα αμήνης, μιλούμε για τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης του AI για να καταγράφει στο λογισμικό κώδικα παράσιτα, επιβλαβή λογισμικό, πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα, πόσο θα αντέξει εφόσον πραγματοποιηθεί επίθεση. Πώς θα ανταποκριθεί επίσης το σύστημα. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να διαμορφώσει αντιμετώπιση αποτελεσματική. Ε, προφανώς επίσης αν έχουμε μια σημαντική υποδομή τηλεπικοινωνιών π.χ. Χρειάζεται συνήθως μήνες ώστε μια ειδική ομάδα τεχνικών να εντοπίσει που βρίσκεται το πρόβλημα. Με την τεχνητή νοημοσύνη κερδίζουμε χρόνο. Γιατί από μήνες μιλούμε πλέον για ώρες. Αυτά είναι τα τρία R καθήκοντα της ε, κυβερνασφάλειας. Και γι' αυτό έχουμε και διάφορες πρωτοβουλίες από την ε, ε, διαταγή των ΗΠΑ ε, για την τεχνητή νοημοσύνη στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη σχετική Cyber Security Act, τις κατευθύνες γραμμές και την έκθεση για την ανάπτυξη προτύπων. Υπάρχει όμως ένα θέμα γιατί όλες αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται στο ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο όψεις θέλουμε να εμπιστευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί έτσι θα εξωθήσουμε την καινοτομία αλλά η εμπιστοσύνη είναι μια περίπλοκη έννοια. Γιατί υποτίθεται ότι μπορείς να αναθέσεις ένα καθήκον αλλά χωρίς να ελέγχεις πώς θα εκτελεστεί αυτό. Μιλούμε λοιπόν για ανάθεση χωρίς έλεγχο. Η αξιοπιστία μπορεί να καταμετρηθεί με δύο τρόπους με την προβλεψιμότητα της συμπεριφορά του φορέα που εκτελεί. Αν έχουμε ένα σύστημα που αγοράζει ένα αγαθό, γάλα, μπορούμε να προβλέψουμε την αξιοπιστία του πόσο αποτελεσματικά το κάνει αυτό. Αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να εκτιμήσουμε ίσως τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του. Γιατί όπως σας έλεγα στην αρχή είναι κλειστό κουτί, είναι black box. Επίσης τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνης είναι ευάλωτα. Έχουμε πάρα πολλέ μελέτες που με ένα μικρό ποσοστό δηλητηριασμού των δεδομένων το σύστημα συμπεριφέρεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Επίσης αν παρέμβει κανείς λίγο με τα ε, μοντέλα κατηγοριοποίησης μπορεί ένα όπλο στα μάτια του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης να φαίνεται λουλούδι και να τροποποιεί επομένω τη συμπεριφορά του. Ένα σήμα stop της τροχιάς μπορεί να δείχνει στο σύστημα σαν σήμα επιτάχυνε αυτό σχετίζεται με τη φύση της απειλής που αντιμετωπίζουμε. Σε προηγούμενες επιθέσεις, αν δούμε εξαγωγή δεδομένων ή παρέμβαση στην ομαλή λειτουργία του συστήματος, ήταν απόπειρε για να αποκτήσει κανείς τον έλεγχο του ίδιου του συστήματος. Έστω ότι ένα σύστημα AI ελέγχει την πρόσβαση σε ένα κτίριο. Αλλά με μία επίθεση, ένας hacker μπορεί να αλλάξει την συμπεριφορά του συστήματος, ώστε να αφήσει μέσα στο κτίριο να επιτρέψει την πρόσβαση στο μόνο άνθρωπο που θέλαμε να του απαγορεύσουμε την πρόσβαση. Το πόσο ισχυρό ή μη ευάλωτο είναι ένα τέτοιο σύστημα το υποστηρίζουν διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες αλλά πρόκειται για μια περίπου ουτοπία για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί ένα σύστημα αυτό να είναι απολύτως ασφαλές σε οποιαδήποτε περίπτωση. οι ανάγκες ενός συστήματος αμυντικού εκτιμώνται και υπολογίζονται, ποσοτικοποιούνται από το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά επειδή είναι κλειστά κουτιά αυτά τα συστήματα, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πότε πήγε κάτι λάθος. Δηλαδή ταυτοποιεί σωστά αυτή τη στιγμή τα malware το σύστημα ή μήπως έχει, υπάρχει κάποια άλλη παγίδα και ταυτοποιεί ως malware κανονικό λογισμικό. Όταν μιλούμε για ε, ε, εύρωστο σύστημα, προσπαθούμε να καταλάβουμε με πόσο διαφορετικό τρόπο μπορεί από την κανονική του συμπεριφορά όταν τροφοδοτείται με δηλητηριώδες λογισμικό πόσο μπορεί να αντέξει, δηλαδή να διατηρήσει την κανονική του συμπεριφορά. Όταν μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη όμως ο αριθμός των δυνητικά δηλητηριωδών λογισμικών δεδομένων πάει μέχρι την ελάχιστη λεπτομέρεια. Μιλούμε για παράδειγμα για ταυτοποίηση προσώπων. Σε επίπεδο πίξελ μπορούμε να τροποποιήσουμε ελάχιστα μια εικόνα. Εάν δεν είναι επαρκώς εύρωστο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, τότε δεν είναι αξιόπιστο. Και αυτό επηρεάζει το θέμα της εμπιστοσύνης. Όταν μιλούμε για οπλικά συστήματα αμήνε, όλα αυτά καθίστανται αρκετά επικίνδυνα σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει λύση. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος φιλόσοφος, λέει ο Μιλήτρια. Πρέπει να μπορούμε να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο χρησιμοποιώντα τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνης για την κυβερνασφάλεια. Καταρχά χρειαζόμαστε ανάπτυξη χωρίς εξωτερική ανάθεση. Μπορεί κανείς να αγοράσει το πρότυπο, το μοντέλο, τα δεδομένα, να τα αναπτύξει. Αλλά έτσι ακριβώς, αυτή είναι η δίωδος από την οποία έρχονται, εισέρχονται και οι επιθέσεις. Αν μιλούμε για την προστασία κρίσιμων υποδομών, πρέπει να αυξήσουμε τα πρότυπα. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις στις οποίες ανατίθεται το οποιοδήποτε καθήκον αρμοδιότητα να έχουν εσωτερική ικανότητα ανάπτυξης. Επίσης υπάρχει μια κατάρτιση, ε, ε, ένα πρόγραμμα δοκιμής όπου βάζουμε δύο συστήματα, το ένα να αντιπαρατεθεί με το άλλο, να συγκρουστεί με το άλλο και μέσω της διαδικασίας αυτής αναπτύσσουμε την, ε, το πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη ή πόσο μπορεί να αντέξει έναντι επιθέσεων. Επίση, πρέπει να αναπτύξουμε πρότυπα όταν χρησιμοποιούμε συστήματα τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο τη άμυνα με έναν, ψηφιακό κλόνο έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε ότι αν ένα σύστημα βρίσκεται εκτός ελεγχόμενου πλαισίου, πότε έχει ξεφύγει από τις παραμέτρους που του έχουμε θέσει. Μιλούμε λοιπόν για μια οντότητα που είναι διαδραστική, αυτόνομη και αυτοδίδακτη. Ή μάλλον αυτοδιδασκόμενη. Το σύστημα μαθαίνει περισσότερα πράγματα, αλλάζει τον εαυτό του και επομένως πρέπει να εντάξουμε πλέον στα αριθμιστικά μας πλαίσια δυναμικό έλεγχο, μεταβλητό έλεγχο. Γιατί ο κίνδυνος θα αλλάζει μαζί με το σύστημα. Και ιδιαίτερα όταν μιλούμε για κρίσιμα αισθήματα μήνης, πρέπει να πάμε από το αξιόπιστο μάλλον από ένα σύστημα που μπορούμε να εμπιστευθούμε σε ένα σύστημα για το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο. Αυτά κάνω με το εργαστήριο στην Οξφόρδη, μερικά από αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Ο Κρίς Πέτερς πρώτος εξ του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους τρεις ομιλητές μας. Είναι προφανές για μένα ότι η όλη αυτή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα πολύπλοκη και βέβαια δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σήμερα. Νομίζω ότι ε, πολλά πράγματα θα χρειαστεί να συζητήσουμε και στο μέλλον για το πώς θα διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, ακούσαμε κάποιες συστάσεις, ορισμένα συμπεράσματα, όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Τώρα, η δική μου ερώτηση είναι η ακόλουθη. Από ό,τι κατάλαβα, οι νέοι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι, Βεστάγκερ και άλλοι, που ανέλαβαν την εντολή τους από την 1η Δεκεμβρίου, δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τις μη στρατιωτικές εφαρμογές της. Και από ό,τι κατάλαβα, προτίθενται να προσπαθήσουν να καλύψουν κάποια οριζόντια ζητήματα, όπως αυτό της διαφάνειας. αλλά λένε όμως ότι θα έχουν εν συνεχεία και μια τομιακή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την κινητικότητα, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και το καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το μη στρατιωτικό σκέλος, ενώ εμείς σήμερα συζητάμε για τη χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας. Εκεί νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να έχει κανείς μια σφαιρική προσέγγιση και ένα κοινό νομικό πλαίσιο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να περιμένουμε να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νομικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης για τις μη στρατιωτικές εφαρμογές, να δούμε δηλαδή τι θα προτείνουν οι αρμόδιοι επίτροποι πρώτα και στη συνέχεια μόνο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τον τομέα της άμυνας γιατί όπως σας είπα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και έπειτα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι, θεωρώ, πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να έχουμε μια γενική συμφωνία για τις πτυχές μη διάδοσης, για παράδειγμα, των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δεν θα έπρεπε όμω να ακολουθήσουμε περισσότερο αυτή τη σειρά, να δημιουργήσουμε πρώτα ένα νομικό πλαίσιο για τον μη στρατιωτικό τομέα και εν συνεχεία να δούμε πώς μπορούμε να πλαισιώσουμε νομικά την τεχνητή νοημοσύνη για τον τομέα της άμυνας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Ρουσλή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω και εγώ για τις πολύ ενδιαφέρουσε αυτές τις παρουσιάσεις. Πολλές παρατηρήσεις και ερωτήσεις θα μπορούσα να κάνω. Πρώτον, προβλέπεται ένας παγκόσμιο παγκόσμιος κανονισμός, διεθνής κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα προβλήματα με τις διεθνείς συμβάσεις, όπως με τη σύμβαση ENF, Όλες αυτές οι απαρελθούσες συμφωνίες για τη μη διάδοση διαφόρων οπλικών συστημάτων βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή καταραίουν. Πώς μπορούμε ποτέ λοιπόν να έχουμε στο μέλλον μια αξιόπιστη διεθνή συμφωνία για τη χρήση της τεχνητής νομοσύνης. Δεύτερον, μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η τεχνητή νομοσύνη αποτελεί κάτι αόριστο που αφορά περισσότερο το μέλλον. Βλέπω όμω τώρα ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Ακόμα και στη Συρία χρησιμοποιούνται εφαρμογέ ρομποτική στον τομέα της άμυνας. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί λοιπόν πραγματικότητα στις εμπόλεμες σειράξεις. Σίγουρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι πλέον θεωρητικό ή φιλοσοφικό. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιτρέψουμε στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να ασχοληθούν, αν θέλετε, με την καταστροφή συγκεκριμένων στόχων, γιατί βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα ήδη γίνονται. Οι αγορές ε, ε, τεχνητής ε, αμυντικού εξοπλισμού και το καθεξής. Θα επιτρέψουμε όμως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο να εντοπίζουν το στόχο, αλλά να πατάνε και το κουμπί για την καταστροφή του στόχου και στους υπόλοιπους στρατούς στην Ρωσία, στις Ηνωμένε Πολιτείε, Ήδη γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται πλήρως και εμπράκτος μάλιστα. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντεμιρέλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω ότι όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη δεν μιλάμε απλώς για καθαρά αυτόνομα οπλικά συστήματα και τι ακριβώς ε, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα αποκλείει, ναι ή όχι. Και πολύ λυπάμαι γιατί βλέπω ότι δεν είναι σαφής εδώ η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον αποκλεισμό. Μιλάμε για ηθικά συστήματα, ηθικούς ε, αλγορίθμους. Πώς είναι δυνατόν ε, το θέμα της ηθικής δεν είναι μόνο θέμα λογικής, αλλά και θέμα συναισθημάτων και συγκινήσεων. Πώς μπορεί κανείς να τα διακρίνει αυτά και πώς μπορεί η απόφαση να εντοπιστεί ένα στόχος και να εξαλειφθεί, να λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από έναν αλγόριθμο. Λυπάμαι πάρα πολύ και κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε εδώ να τοποθετηθούμε σαφώς υπέρ μιας απαγόρευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πάρουν μια τέτοια θέση, ότι δηλαδή τα αυτόματα αυτά συστήματα, τα φωνικά και τα οπλικά, είναι ακριβώς την ίδια κατηγορία όπως και τα πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να απαγορευτούν κύριος Νταμιτζά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Ταντέο συνόψισε πάρα πολύ καλά την όλη συζήτηση, η τελευταία μιλήτρια δηλαδή. Δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς τα συστήματα αυτά ακόμα εντελώς αξιόπιστα, αλλά αν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά, μπορούμε να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Να σας δώσω το παράδειγμα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, του, της Τέσλα για παράδειγμα, όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς ε, την αυτόματη οδήγηση και χρησιμοποιεί μόνο GPS. Αυτή τη στιγμή εσείς εκεί ως οδηγός και παρακολουθείς την κατάσταση έχει καλώς. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή τη στιγμή ε, όλοι συνηθίσουν να χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα, αυτό τα πράγματα θα αλλάξουν συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τον τομέα της άμυνας από ότι με τις υπόλοιπες μη στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, λέει Πρόεδρος, να θέσω κάποιες ερωτήσεις που ουσιαστικά αποτελούν συνέχεια των όσων είπαν μόλις τώρα οι συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να είχα μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του επίπεδου χρησιμοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης ιδίως των αυτόνομων συστημάτων, των αυτόνομων φωνικών οπλικών συστημάτων στον αμυντικό εξοπλισμό χωρών όπως η Ρωσία και η Κίνα ή ακόμα και η Βόρεια Κορέα. Αναφερόμαστε σε κάτι υποθετικό αυτή τη στιγμή, σε εικασίες ή υπάρχει όντω η χρησιμοποίηση αυτή από τι χώρε αυτέ. Επίση, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σα για ένα άλλο ζήτημα σε ποιο βαθμό τα φωνικά αυτόνομα οπλικά συστήματα σήμερα ή στο εγγύς μέλλον μπορούν να πέσουν στα χέρια μη κρατικών φορέων ενδεχομένως. Και στην περίπτωση αυτή να χρειαστούν οι δικές μας οι ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιστάσεις. Και σε επιχειρήσεις βέβαια και αποστολές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα μία ερώτηση ανθρώπου που δεν είναι ειδήμων. Ποιο είναι το ζήτημα της τιμής του κόστους όσον αφορά αυτά τα φωνικά αυτόνομα οπλικά συστήματα. Είναι συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι πιο πλούσιες χώρες και άρα θα μιλάμε για ένα πόλεμο πλουσίων εναντίον των φτωχών η διάδοση των οπλικών αυτών συστημάτων ενδεχομένω να οδηγήσει τελικά σε μια εύκολη προσβασιμότητα στα όπλα αυτά από πάρα πολλούς φορείς και όπως σας είπα και από μη κρατικούς φορείς τελικά. Και εν τέλει και σε σχέση με ένα ερώτημα το οποίο ακούσαμε στο υφιστάμενο πλαίσιο όλων αυτών των ε, διεθνών προσπαθειών ελέγχου των ε, εξοπλισμών των αμυντικών, που όπως είπαμε οι συμβάσεις αυτές όλο και περισσότερο τελικά δεν τηρούνται από κάποιες ε, μεγάλες δυνάμεις, σε ποιο βαθμό οι όλες οι συζητήσεις που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν πραγματικά να σημειώσουν πρόοδο και ποια είναι η άποψη που εκφράζουν κυρίως οι μη ευρωπαϊκοί φορείς στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Maybe uh, I will start on... Να ξεκινήσω, Πρόεδρε, με κάποια από τα θέματα αυτά, όχι όλα ίσως. Έγινε μια ερώτηση ε, πόσο πρέπει να περιμένουμε στο πολιτικό πλαίσιο. Νομίζω ότι το πολιτικό με το στρατιωτικό πρέπει να εξελιχθούν παραλλήλως. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε ούτε στα θέματα αμήνης. Κάποιες στοιχείες βεβαίως διαφοροποιούνται. Αυτά που σχεδιάζονται για την προστασία των καταναλωτών ή των πολιτών, των πολιτών με την έννοια του καταναλωτή, λέει ο μιλητή ακριβώς, πρέπει να το δούμε διαφορετικά στο επίπεδο της αμήνης. Υπάρχουν θέματα ιδιωτικότητας, τα οποία συνδέονται αλλά όχι υποχρεωτικά με την άμυνα. Σε γενικές γραμμές αυτό που θα προσέφερε προστιθέμενη αξία θα ήταν να μπορούμε να δοκιμάζουμε μια λύση τεχνητής νοημοσύνης ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον σε ερευνητικό επίπεδο τι κάνουν οι αλγόριθμοι και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε, να διατηρούμε τον έλεγχο του συστήματος και να κινηθούμε προς αυτό το θέμα αξιοπιστίας κάθετος εμπιστοσύνης, του οποίου η μεθόριος ε, είναι αρκετά συγκεχημένη για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή πλήρως αυτόνομων συστημάτων μάλλον αυτό μάλλον στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ των δύο της Βορείου και της Νοτιού Κορέας μάλλον ε, είναι ήδη ανεπτυγμένα αυτόνομα συστήματα. Τώρα, υπό την έννοια του λογισμικού, Μιλούμε για μια ψηφιακή τεχνολογία και ε, έχει αν θέλετε μια τάση εκδημοκρατισμού. Δηλαδή επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες πρόσβαση. Και οπωσδήποτε και μη κρατικοί φορείς θα χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες. Θα είναι πιο δύσκολο να ρυθμίσει, να ελέγξει κανείς την τεχνολογία αυτή και θα πρέπει σίγουρα να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και στα θέματα της ε, αμυντικής ε, τεχνολογίας. Ε, συμφωνώ και εγώ, Πρόεδρε, με πολλούς από τους ομιλητές και τις ερωτήσεις. Ε, τα αυτόνομα συστήματα ήδη υφίστανται. Πέρα από τα οπλικά συστήματα Sentry που ανέφερε ο συνάδελφος, έχουμε επιθετικά οπλικά συστήματα που μπορεί κανείς, ας πούμε, να αναπτύξει στον αέρα ε, για παράδειγμα κινητός εκτοξευτής πυράβλων. Δηλαδή ήδη υπάρχουν αυτά τα συστήματα, χρησιμοποιούνται. Έχουμε βεβαίω πολύ μεγάλη ποικιλία, διαφοροποίηση. Ε, ίσως κάποια να μην είναι τόσο τελειοποιημένα, αλλά θα μπορούσαν να τελειοποιηθούν στο μέλλον και να επιτύχουν ε, πολύ καλύτερη, καλύτερες επιδόσεις. Επίσης το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά θα ήταν λάθος να κοιτούμε απλώς το θέμα των φωνικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων όπου ο άνθρωπος λαμβάνει την τελική απόφαση. Εδώ μιλούμε για μια σταδιακή βραδία εκρίζωση τη συμμετοχή του ανθρώπινου φορέα. Ε, πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση ε, για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι άνθρωποι σε πλαίσια στόχευσης, σε συστήματα στόχευσης. Ίσως ε, να πολλαπλασιαστούν συστήματα πιο απλά, επιθετικά, σε μη κρατικούς φορούς, φορείς, με συγχωρείτε, με δεδομένα που θα βρίσκουν στο διαδίκτυο. Σίγουρα μη κρατικοί φορείς θα μπορέσουν να αποκτήσουν τέτοια συστήματα. Επίσης μιλούμε συχνά για τους εσμούς, για την τεχνολογία των swarms. Ένας εσμός, μια ομάδα στοιχείων που λειτουργεί ως ενιαία οντότητα είναι κάτι που σίγουρα θα δούμε. Επίσης μιλούμε για το πόσο υλοποιήσιμα είναι αυτά τα συστήματα. Η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Κίνα ειδικά είναι αφενός μας λέει ότι εναντιώνεται στην νομοθετική αυτή δραστηριότητα. Από την άλλη μιλάει για πάρα πολύ υψηλά πρότυπα και ε, ευφυΐα ε, ισότιμη με την ανθρώπινη. Είναι λίγο δύσκολο να καθορίσει κανείς την τοποθέτησή της. Το γεγονό ότι είναι δύσκολο δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσουμε και το ίδιο ισχύει για τα πυρηνικά όπλα που είπατε. Είναι πολύ δύσκολο το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά ιδιαίτερα αυτό και ιδιαίτερα σε περιοχέ υψηλή ένταση όπω σήμερα, μα χρειάζεται αυτό και πρέπει να διέπει τη σχέση μεταξύ των χωρών. Η κυρία Ταντέο. Δύο νομίζω σημεία έχω μόνο. Το πρώτο, μετά από και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, το γεγονός ότι είναι δύσκολο να νομοθετήσουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσουμε. Έχουμε κάνει και πιο δύσκολα πράγματα ως είδος στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει και άλλη όψη στο νόμισμα. Εστιαζόμαστε ιδιαίτερα στα φωνικά αυτόνομα συστήματα και ξεχνούμε υφιστάμενες εκφάνσεις της τεχνητής νοημοσύνης που είναι ιδιαίτερα καταστροφικές και καθόλου ελεγχόμενες. Όσο δεν είναι κινητικά αυτά τα συστήματα, δεν ρυθμίζονται, δεν νομοθετούνται. Δεν χρειαζόμαστε δεν είναι πλέον το πρόβλημα ότι πρέπει να, να μην χρησιμοποιήσουμε την ατομική βόμβα. Μιλούμε για κρίσιμε υποδομέ και απλέ. Νοσοκομεία, δρόμου. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλή στο να επιτίθεται σε τέτοια υποδομή. Και αυτά θα διαχυθούν ακόμα πιο έντονα από τα φωνικά αυτόνομα στήματα τα οποία προϋποθέτουν και σημαντικούς πόρους. το κακόβουλο λογισμικό ενός συστήματος τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη διαθέσιμο. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Και εδώ έχουμε κρατικούς φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο αυτό. Θα ήταν δύσκολο ενδεχομένως να έχουμε έναν παγκόσμιο κανονισμό, ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά έχουμε άλλα εργαλεία. Τυποποίηση, συμμαχίες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να μην έχουμε συμμαχίε μεταξύ χωρών για, για συστήματα ε, ε, αντιμετώπισης κρίσιμων κενών. Το UNACRA, για παράδειγμα, ήταν μια ε, ε, χαρακτηριστική περίπτωση γιατί να μην μπορούμε να συνεργαστούμε για να νομοθετήσουμε ή να ρυθμίσουμε τις πτυχές εκείνες που σχετίζονται τουλάχιστον με στρατιωτικές συμμεχίες πώς μια συμμαχία μπορεί να είναι πιο συντονισμένη και πιο αποτελεσματική ως προς αυτό. Για το αν πρέπει η εστίασή μας να είναι στα πολιτικά ή στα στρατιωτικά στήματα θα έλεγα να το αποφύγουμε αυτό το διαδικό. Η απειλή είναι ήδη εδώ. Δεν θέλω τώρα να εμφανίζουμε εδώ ως πανδώρα, αλλά ε, έχουμε απειλές για τις πολιτικές υποδομές. και θα έχουμε πολύ σημαντικούς κινδύνους και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ όλους όσους πήραν το λόγο και μας παρουσίασαν αυτά τα πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία και προτάσεις. Αυτές οι νέες τεχνολογίες μας προτείνουν και ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά και πραγματικές ε, απειλές και κινδύνους και μπορεί να αλλάξει η φύση, αν θέλετε, της ε, πολεμικής τέχνης. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε, θεωρητική. Ακούσαμε πραγματικές ε, ιδέες και ενδεχομένως αυτό που θέλω να εκφράσω σαν αρνητικό είναι ότι σήμερα δεν μπορέσαμε να ακούσουμε με ξεκάθαρο τρόπο από το μέρος των ειδικών ποια μπορεί να είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο των επιχειρήσεων. Εάν δηλαδή βοηθούν αυτές οι τεχνολογίες και κατά πόσο τους προστατεύουν, τους στηρίζουν στη λήψη αποφάσεων και κατά πόσο τους ανησυχούν. Μας περιγράψατε, η τελευταία ομιλήτρια περιέγραψε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ευάλωτη σε παρεμβάσεις, σε επιθέσεις και πώς αυτά τα αυτόμα, αυτόνομα συγγνώμη, οπλικά συστήματα ε, μπορεί να επηρεάσουν την πραγματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως συνήθως ε, θα συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτού του θέματος με την ε, Επιτροπή μας αλλά και με άλλες. Θέλουμε πραγματικά να δείξουμε ότι ότι και εμείς ε, λειτουργούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές. Θα ξαναρχίσουμε στις 2.30 το απόγευμα.